We start meeting. Uh, all the languages are available. Αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός από κροατικά και μαλτέζικα. Έχουμε κάποιες αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής μας. Ο κύριος Τόμ Φαντεν Κέντελα είναι αναδροματικό μέλος της Επιτροπής μας από πλευράς του ΕΛΚ. Είστε παρόν. Α, καλώς ήρθατε. Η κυρία Κορίνα Κρέτου ορίστηκε επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική. Δεν είναι λοιπόν πλέον μέλος της Επιτροπής μας, ούτε του Κοινοβουλίου. Επειδή η κυρία Βέμπερ πήγε από το ΕΛΚ στο ΑΛΔΕ, το ΕΛΚ έχει 15 θέσεις στην Επιτροπή μας αντί για 16 και η Άλντε θα λάβει μία έκτη. Μέχρι στιγμής είχαν πέντε. Yes. Uh, I think... Και ήδη έχουμε τον αντικαταστάτη της κυρίας Κρέτου, είναι ο κύριος Πάβελ. Ε, ε, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις. Τώρα κάποιες συνεδριάσεις που θα κάνουμε. μπορείτε να βάλετε στο ημερολόγιο σας την κοινή συνεδρίαση Econ ΕΜΠΛ για την ετήσια μελέτη για την ανάπτυξη. Θα γίνει στις 2 12 από τις 8 έως τις 10 σημαντική συνεδρίαση και κατόπιν στην ίδια αίθουσα Γιάν 4Q2 θα έχουμε μία ακρόαση για το TTIP που επίσης είχαμε ζητήσει να διεξαχθεί και η οποία θα αρχίσει στις 10 αλλά στην αίθουσα που είμαστε τώρα PHS 3 σε 50 Δύο λοιπόν σημαντικές ε, συνεδριάσεις για την Επιτροπή μας Έχουμε αυτή τη συνεδρίαση λοιπόν για την ετήσια μελέτη για την ανάπτυξη και μετά για το TTIP. Δύο λοιπόν διαδοχικές ακροάσεις. Επίσης, στη συνέχεια θα δώσουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για την Νεότητα που διεξήχθη τον Μάιο στο Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Ως συνέχεια αυτής της εκδήλωσης θα έχουμε μια άτυπη εκδήλωση θα έχουμε μια ειδική διαδικασία που λέγεται εξακρίβωση ιδεών θα έχουμε 60 λεπτά συνεδρίασης κατά την οποία οι νέοι θα είναι αυτοί που θα κάνουν προτάσεις για ιδέες και εμείς θα είμαστε ως μέλη του Κοινοβουλίου οι αποδέκτες του. Δηλαδή θα κληθείτε να σχολιάσετε απευθείας τις ιδέες που θα προτείνουν οι νέοι. Και ελπίζω να έρθετε πολύ. Δεν είναι δυνατόν να καλέσουμε τους νέους, να τους φιλοξενήσουμε λίγο πριν τις εκλογές και μετά να μην ασχοληθούμε μαζί τους και με τις ιδέες τους λίγους μήνες αργότερα. Ελπίζω λοιπόν να προσέλθετε σε αυτή τη συνεδρία σε αυτή την ειδική ταχυακρόαση. Έγκριση των πρακτικών. Υποθέτω δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο ψηφοφορία. Παρακαλώ να έχετε τις κάρτες σας. I hope managed. We have to... Εντάξει. Ωραία. Πρέπει να ελέγξουμε εφόσον, ε, εφόσον πρόκειται να ψηφίσουμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Έχουμε δύο θέματα. Το πρώτο είναι η κινητοποίηση του ταμείου αυτού για την ε, περίπτωση Whirlpool στην Ιταλία. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Πέρας. Πέρας. Ωραία. Τώρα να ψηφίσουμε για την ε, κινητοποίηση του Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Α, δεν ανακοίνωσα το αποτέλεσμα. Α, μάλιστα. 32 υπέρ. 3 κατά. και καμία αποχή. Επόμενη ψηφοφορία. Μπορούμε να δούμε τα... το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Ωραία. Επαναλαμβάνει την ψηφοφορία. Πέρας. Έχουμε και μία αποχή. 3 κατά, 33 υπέρ. Τώρα να, να ψηφίσουμε για το δεύτερο θέμα. Πάλι η κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση για την γαλλική περίπτωση της εταιρείας GAD. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 34 υπέρ, 3 κατά και 1 αποχή. Ευχαριστώ πολύ. Now we'll have the report from the Commission on the... Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 104 2008 για την εργασία των ε, εταιριών προσωρινής απασχόλησης και να δώσω το λόγο στον κύριο Αρμίντα Σίλβα από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Είναι η Διευθυντής για την Απασχόληση και την Κοινωνική Νομοθεσία και έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. να σας παρουσιάσω πρώτα απ' όλα το πλαίσιο και το περιεχόμενο της οδηγίας 2008 κάθετος 104 για την εργασία μέσω εταιρεών προσωρινής απασχόλησης και θα παρουσιάσω και τα κύρια πορίσματα της έκθεσης που δημοσιεύθηκε τον παρελθόντα Μάρτιο και θα πω και ορισμένα λόγια για το τι συνέχεια θα δώσουμε στην οδηγία. Η οδηγία αυτή λοιπόν αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται μέσω μιας εταιρείας προσωρινής απασχόλησης. ΕΠΑ. Για να αξιοποιηθούν από έναν εργοδότη υπό την επίβλεψη και καθοδήγησή του. Έχουμε λοιπόν μια τριμερή σχέση. Τον ε, εργαζόμενο, τον εργοδότη και την εταιρεία αυτή. Αυτή είναι μια όχι συνηθισμένη μορφή απασχόληση που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε ότι 1,6% του εργατικού δυναμικού της Ένωσης εργάζεται με αυτό το είδος εργασίας. Πολύ υψηλέ διακυμάνσεις ανά χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία έχουν πολύ ψηλότερο ποσοστό. Και βεβαίως αυτού του τύπου απασχόληση επηρεάζεται πολύ από τον οικονομικό κύκλο. Αυτός ο τύπος εργασίας είναι πολύ ευέλικτος για τις εταιρείε, τους προσφέρει ευελιξία και μπορεί να είναι και ένα σκαλοπάτι προς μια πιο μόνιμη απασχόληση για τους ανέργους. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι επισφαλής. Η οδηγία αυτή έχει μακρά ιστορία. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, η Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, οι οποίες απέτυχαν το 2001 και μετά το 2002 η Επιτροπή αποφάσισε να κάνει προτάσεις οδηγίες που χρειάστηκαν 6 χρόνια διαπραγματεύσεων, κυρίως στο Συμβούλιο και η κύρια δυσχέρεια αφορούσε τις εξαιρέσεις από την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Όπως θα πω περαιτέρω. Στόχος της οδηγίας όπως τελικά εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ήταν πρώτον να βελτιωθεί η προστασία των εργαζομένων αυτού του τύπου μέσω της ε, εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Αλλά παράλληλα να αναγνωρίσει και να στηρίξει το θετικό ρόλο αυτής της μορφής εργασίας και των εταιριών ΕΠΑ στην ε, εισαγωγή ευελιξίας στην αγορά εργασίας μέσω απάλληψης ε, των ε, υπερβολικών περιορισμών. Στα πρώτα άρθρα καθορίζουμε την ίση μεταχείριση. Είναι μία αρχή που θα πρέπει να ισχύει για όλους αυτούς τους εργαζόμενους για τις βασικές σχέσεις απασχόλησης και εργασίας, δηλαδή την αμοιβή και το χρόνο εργασίας. Στο άρθρο 5 καθορίζουμε κάποιες ε, περιορισμένες εξαιρέσεις υπό αυστηρές συνθήκες. Τρεις σημαντικές εξαιρέσεις. Πρώτη, στην παράγραφο 2, αφορά τους εργαζόμενους που έχουν μόνιμο συμβούλιο. Έχουν δηλαδή αορίστου χρόνου ε, και πληρώνονται και όταν δεν εργάζονται. Αυτό θεωρείται βασικό πλεονέκτημα που επιτρέπει να μην υπάρχει ίση αμοιβή. Και στην τρίτη παράγραφο εισάγουμε τις εξαιρέσεις μεταξύ συλλογικών συμφωνιών. Εάν υπάρχουν συλλογικές συμφωνίες μπορούν να θεσμοθετούν εξαιρέσεις. Και τέλος, και αυτό ήταν το πιο δυσχερές σημείο στο Συμβούλιο, χρειαστήκαμε χρόνια για να καταλήξουμε, στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 λέμε ότι τα κράτη-μέλη που δεν έχουν σύστημα για την επέκταση, για την επιμήκυνση των συλλογικών συμβάσεων ή κανένα σύστημα συλλογικών ε, συμφωνιών, τους δίνουμε δυνατότητα όχι μόνο να κάνουν εξαιρέσεις, αλλά και να εισαγάγουν μία ε, μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης μετά από συμφωνία σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Και το άρθρο 4 είναι σημαντικό της οδηγίας ε, όπου θεσμοθετείται υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να αναθεωρούν όλες, όλους τους περιορισμούς και απαγορεύσεις για τη χρήση της εργασίας αυτής και τονίζει ότι περιοριστικά μέτρα μπορούν να αιτιολογηθούν μόνο για λόγους γενικού συμφέροντος. Για παράδειγμα, η προστασία των εργαζομένων, της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας και η σωστή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Δημιουργεί υποχρέωση για τα κράτη-μέλη την οποία πρέπει να τηρούν και να στέλνουν και εκθέσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έπρεπε να έχουν στείλει εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2011. Σημαντικό και το άρθρο 6, οι εργαζόμενοι αυτοί, μέσω αυτού του άρθρου έχουν τη δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης στην ε, μόνιμη εργασία. Και το άρθρο 7 καθορίζει τους όρους εκπροσώπησης των εργαζομένων αυτών και την ενημέρωση των εκπροσώπων τους. Είτε σε αυτές τις ε, ειδικέ εταιρείες Η οδηγία δημιουργεί για την Επιτροπή την υποχρέωση να αναθεωρήσει την εφαρμογή της οδηγίας, να εξετάσει μάλλον την εφαρμογή της οδηγίας και να υποβάλει έκθεση με στόχο, εάν χρειάζεται, να προταθεί η τροποποίησή της. Η έκθεση αυτή λοιπόν εκπονήθηκε σε στενή διαβούλευση με τα κράτη-μέλη και τους ε, κοινωνικούς εταίρους. Υπάρχει μια επιτροπή που ιδρύθηκε από αυτή την έκθεση με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των κρατών μελών. Ακούσαμε και εμπειρογνώμονες και τελικά δημοσιεύσαμε αυτή την έκθεση τον παρελθόντα Μάρτιο, όπως ε, ήδη είπα. Η έκθεση αυτή έχει και παραρτήματα τεχνικού τύπου. Βλέπετε εδώ τα slide. Τι λέει η έκθεση κυρίως, ποια είναι τα κύρια πορίσματα. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν την οδηγία. Ορισμένα κράτη-μέλη το έκαναν με πολύ καθυστέρηση. Δεν έχουμε πολλή εμπειρία από την εφαρμογή της. Πρέπει να το έχουμε λοιπόν υπόψη γιατί η περίοδος μεταγραφής έπρεπε να έχει λήξει το 2011. Ορισμένα κράτη-μέλη όμως καθυστέρησαν και την μετέγραψαν το 2012 οπότε έχει εφαρμοστεί για λίγο. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα όπου δεν είδαμε ιδιαίτερες δυσχέρειες εφαρμογής, πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, πρόσβαση στην απασχόληση, συλλογικές ε, ε, εγκαταστάσεις, εκπροσώπηση των εργαζομένων. Δεν ε, διαπιστώσαμε δυσχέρειες για την εφαρμογή αυτών των στοιχείων. Για τις εξαιρέσεις από την αρχή της ίσης μεταχείρισης, σε 12 κράτη-μέλη διαπιστώσαμε κάποια μορφής εξαιρέσεις. Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μόλτα, Μάλτα, Ολλανδία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Για το άρθρο 4, η εξέταση των περιορισμών και απαγορεύσεων, όλα τα κράτη-μέλη ενημέρωσαν την Κομισιόν για τα αποτελέσματα της δικής τους εξέτασης. Μόνο ένα κράτος μέλος δεν το έχει πράξει. Τρία κράτη-μέλη θεωρούν ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί. Και η έκθεση αναφέρει τις κύριες αιτιολογήσεις για αυτούς τους περιορισμούς και ποια διαβούλευση έγινε με τους κοινωνικούς εταίρους. Τώρα το κόστος για τις ρυθμιστικές διατάξεις. Είχαμε μια ειδική έρευνα γι' αυτό δεν είχαμε παράπονα από τις αρχές των κρατών μελών για ουσιώδες συμπληρωματικό κόστος λόγω της εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Αλλά, κατά την άποψη των εργοδοτών, οι περιορισμοί στην ε, δραστηριότητα των ΕΠΑ δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς από τις εθνικές αρχές. Και ορισμένοι από αυτούς τους περιορισμούς συνεχίζουν να έχουν ως συνέπεια κόστος για την οικονομία. Ορίσματα λοιπόν της ε, έκθεσης αυτής, γενικά, θεωρούμε ότι η οδηγία έχει εφαρμοστεί σωστά. Όμως από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής ο διτός στόχος οδηγίας τον οποίον ήδη ανέφερα δεν έχει επιτευχθεί πλήρως. Πρώτον, η αρχή της εις Αναγνωρίζουμε ότι η χρήση κάποιων εξαιρέσεων και κάποιες ερμηνείες από κάποιες εθνικές αρχές για το πώς πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι οδηγίες μπορεί να πάνε τόσο μακριά ούτω ώστε να μην υπάρχει καμία βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων αυτού του τύπου. Άρα οι εργαζόμενοι αυτοί δεν προστατεύονται στην ουσία και δεν εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τώρα η εξέταση των περιορισμών και απαγορεύσεων αναγνωρίζουμε ότι σε μια σειρά από περιπτώσεις τα κράτη-μέλη αξιοποίησαν αυτή τη ρήτρα για να νομοποιήσουν το status quo χωρίς να εξετάσουν σε βάθος τη σχέση κόστους αποτελέσματος αυτών των περιορισμών. Ωστόσο κάποιοι περιορισμοί καταργήθηκαν λόγω αυτής της ε, εξέτασης του 2011 και θεωρούμε ότι θα υπάρξει περαιτέρω πρόοδος σε κάποια κράτη-μέλη στο θέμα της εξέτασης κάποιων υπερβαλλικών περιορισμών δραστηριότητας αυτών των ε, ΕΠΑ. Η οδηγία αυτή βεβαίως είναι ακόμη σε φάση εφαρμογής. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει την κατάσταση όπως ήταν το τέλος του 2013. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή της. Έχουμε μια επιτροπή όπου συμμετέχουν τα κράτη-μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι. Είναι ένα βήμα διαλόγου που μας επιτρέπει να καθορίσουμε τα προβλήματα. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε δύο μέσα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε τις ε, διαδικασίες επί παραβάση αν θεωρήσουμε ότι κάποια οδηγία παραβιάζεται σε σημαντικό βαθμό. Και αν χρειαστεί θα εφαρμόσουμε αυτή τη δυνατότητα. Και η δεύτερη δυνατότητα είναι οι συστάσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εάν λοιπόν βρούμε ότι υπάρχει υπερβολική ρυθμιστική επιβάρυνση σε κάποιο κράτος μέλος που είναι εμπόδιο για την ανάπτυξη και για την ευέλικτη λειτουργία της αγοράς εργασίας, τότε η Κομισιόν μπορεί να κάνει συγκεκριμένες συστάσεις για τη χώρα. Σε αυτή τη φάση δεν προτιθέμεθα να τροποποιήσουμε την οδηγία. Η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την ορθή εφαρμογή της. Έχουμε ξεκινήσει και λαμβάνουμε κάποια παράπονα, ενστάσεις, καταγγελίες από πολίτες και οργανώσεις, όχι πολλά. Τρεις νομίζω περιπτώσεις έχουμε στους φακέλους μας ε, και τις οποίες και αναλύουμε. Έχουμε και ένα σημαντικό προκαταρκτικό ερώτημα προς το δικαστήριο. Πρόκειται για μια υπόθεση που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από το Δικαστήριο της Φινλανδίας F523 σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του άρθρου 4 Ο καταγγέλων θεωρεί ότι οι εθνικές αρχές δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αναθεωρήσουν και να εξετάσουν τους περιορισμούς. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τις συνέπειες του άρθρου 4 της οδηγίας και παρακολουθούμε το θέμα αυτό επισταμένως καθότι μπορεί να δημιουργηθεί σχετική νομολογία και κατά σύμπτωση σήμερα θα ακούσουμε ποιες ε, είναι, ποια θα είναι τα πορίσματα του Γενικού Εισαγγελέα. Θα έχουμε λοιπόν τα αποτελέσματα σε κάποιους μήνες. Αυτά λοιπόν είχα να σας παρουσιάσω και ασφαλώς ε, με χαρά μου θα απαντήσω ενδεχόμενες ερωτήσεις που έχετε για την έκθεση αυτή. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Σίλβα, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα έχετε το λόγο αν θέλετε για ερωτήσεις. Κύριε Μόγαν Σαχτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σίλβα. Ήταν πληρέστατη η παρουσίαση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας. Έχω κάποια συμπληρωματικά ερωτήματα. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψή σας. Πρώτον, είπατε πως ο στόχος της οδηγίας είναι αυτοί που προσωρινά απασχολούνται να κάνουν ένα βήμα, να ανέβουν ένα σκαλοπάτι που θα τους οδηγήσει σε μία μόνιμη σύμβαση μέσω αυτών των εταιριών προσωρινής απασχόλησης. Έτσι έχουν μία καλύτερη πρόσβαση σε μόνιμες θέσεις εργασίας, αορίες του χρόνου και μόνιμες. Πώς αντιλαμβάνεστε αυτή τη μετάβαση των εργαζομένων από προσωρινή σε μόνιμη επασχόληση. Ενώ βιώνουμε αυτή την οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Ενώ ότι η περίοδος εφαρμογής είναι ε, πάρα πολύ προβληματική λόγω της κρίσης. Πώς μπορεί να υλοποιηθεί ο στόχος. Δεύτερο ερώτημα. Αυτές οι αποκλείς εξαιρέσεις, οποίες αναφερθήκατε, υπάρχει τρόπος να τις μειώσουμε και πώς. Τρίτον, από πλευράς εργοδότη, έχετε αναλύσει αυτό το συμπληρωματικό κόστος που καταγγέλουν για την οικονομία. Και τέταρτον, Ξέρουμε ότι είναι επισφαλέστερες ακόμη θέσεις εργασίας για τις γυναίκες λόγω της κρίσης. Με τις παρατηρήσεις που κάνατε στον τομέα των ΕΠΑ, έχετε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, δηλαδή ανάλυση επιπτώσεων για τις γυναίκες και τους άντρες ξεχωριστά στο πλαίσιο των ΕΠΑ. Θα ήθελα για αυτά τα τέσσερα ερωτήματα να με διαφωτίσετε, είναι Θέλετε να απαντήσετε, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Ναι, μπορώ να απαντήσω ήδη σε αυτό το σετ ε, ερωτήσεων. Ο πρωταρχικός στόχος της οδηγίας, θα ήθελα να επισημάνω, είναι να κατοχυρωθεί η ισότιμη μεταχείριση. Βάσει μιας ρήτρας υπάρχει προνομιακή πρόσβαση ε, στην, ε, ε, στον έμεσο εργοδότη για αυτόν τον εργαζόμενο που αποσχολείται μέσω ΕΠΑ. Δηλαδή, Υπάρχει ειδική ρήτρα στη σύμβαση μετά τη λήξη της προσωρινής σύμβασης πρόβλεψη για μόνιμη απασχόληση. Αυτό είναι ένα παράλληλο, ένα συνοδευτικό μέτρο. Έγινε μια αξιολόγηση οικονομικού αντικτύπου για το ρόλο αυτών των συμβάσεων ως γέφυρα προς συμβάσεις μόνιμης απασχόλησης Μάλλον δεν έχει γίνει ε, μελέτη οικονομικού αντικτύπου, έχουν γίνει διαφορετικού είδους μελέτες που αναλύουν τον οικονομικό κύκλο. Βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτών που πέρασαν από προσωρινή σε μόνιμη απασχόληση, αν θυμάμαι καλά, ανέρχεται σε ε, κάτω του 50% ε, των συμβάσεων. Είναι περιορισμένο το ποσοστό, αλλά ξαναλέω ότι ε, αυτή η μελέτη φέρει επί τις οδηγίες και δεν είναι γενικότερου χαρακτήρα. Δεν έχουμε ε, την πρόθεση να περιορίσουμε τις εξαιρέσεις αποκλήσεις ε, στην οδηγία. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι περιπτώσεις κατάχρησης και, μη, ε, και δυσανάλογης χρήσης αυτών των εξαιρέσεων. αφαιρώντας έτσι προστατευτικά για τους εργαζόμενους μέσα Ε, χαμηλότερη αμοιβή κατά 50% ε, αν συγκρίνουμε δηλαδή ε, μια σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου. Ε, αυτή περίπτωση μπορούμε να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο κάποιος προσφεύγει σε αυτή την εξαίρεση. Κατά περίπτωση όμως θα το κρίνουμε αυτό και επί τη βάση των ε, καταγγελιών που λαμβάνουμε από τις ενώσεις πολιτών ή στα πλαίσια του διαλόγου με τα κράτη-μέλη. Ποιος είναι ο αντίκτυπος στην οικονομία, με ρωτήσατε. Κάναμε έρευνα και στις αρμόδιες εθνικές αρχές και στους εργοδότες. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν μας μίλησαν για υπερβολικό διοικητικό άκθος, υπερβολικό δυσανάλογο διοικητικό κόστος σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας. Οι εργοδότες από την πλευρά τους παραπονέθηκαν για κάποιες ρήτρε της οδηγίας, κυρίως σε σχέση με τη ρήτρα για την ισότιμη μεταχείριση, αλλά και κυρίως για την επιβολή αυτών ε, των περιορισμών που ισχύουν βάσει της οδηγίας και πώς τις χειρίζονται τα κράτη-μέλη. Στα πλαίσια της άσκησης που ονομάζουμε εμείς top 10, δηλαδή σε διοικητικό και ρυθμιστικό πλαίσιο προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε μειονεκτήματα σε επίπεδο επιχείρησης και εκεί ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, παραπονέθηκαν για διοικητικό και ρυθμιστικό άχθος και κόστος ε, με την εφαρμογή της οδηγίας. Δεν μπορούμε όμως να σας δώσουμε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία γιατί η μελέτη δεν έχει γίνει. Πρόκειται όμως ε, κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εγγράφεται αυτό στο πλαίσιο της άσκησης top 10. Ε, ποσοτικοποιημένα και ουσιαστικά στοιχεία δεν έχουμε να σας δώσουμε όμως. Για τις επιπτώσεις για τις γυναίκες. Δεν νομίζω να έχει διεξαχθεί δική μελέτη. Όχι στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ, κύριος Σάιμον. Thank you. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σίλβα για την παρουσίασή σας και για τις επεξηγήσεις που δώσατε. Αναφερθήκατε μερικές φορές στις καταγγελίες που έχετε λάβει από πολίτες και οργανώσεις είπατε και αναφέρατε ότι πρόκειται μόνο για τρεις. Περίεργο περιλαμβάνεται σε αυτές τις τρεις ε, η καταγγελία ε, που υποβλήθηκε στις 3 ε, Σεπτεμβρίου 2013 από το Βρετανικό Συνδικάτο. Πάνω από ένας χρόνος έχει περάσει. Είναι μεγαλύτερη χρονική περίοδο από αυτή που έχει ω προθεσμία Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει σε καταγγελίε. 15 μήνε. Νομίζω ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η βάση τη καταγγελία είναι πάρα πολύ απλή και περιλαμβάνεται στην παρουσίασή σα, η οποία και αναφέρει ότι πρόκειται, ότι πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί αρκετά καλά, εκτός από κάποιες χώρες που χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν παρακλήσεις, όπου σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργεί καθόλου το σύστημα. Το συνδικάτο TUC αναφέρει ότι η παρέκκληση που εφαρμόζεται στον Ομένο Βασίλειο οδηγεί στη μη εφαρμόγη της νομοθεσίας αυτής ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο με επιτυχή τρόπο. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία κατά της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και το έχει, την έχει καταθέσει η βασική οργάνωση εκπροσώπησης εργαζομένων. Πριν από 15 μήνες, επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας παρακαλώ λοιπόν, για πείτε μας ε, λίγα λόγια για την καταγγελία αυτή. Και δώστε μας, ακόμα πιο σημαντικό αυτό, μια ημερομηνία κατά την οποία το Συνδικάτο TUC μπορεί να αναμένει απάντηση σε ό,τι αφορά την ε, εκμετάλλευση τόσων πολλών εργαζομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο από ένα θέμα το οποίο ακριβώς και αποσκοπεί η νομοθεσία αυτή, η απάντηση. Ναι. Να σας επιβεβαιώσω ότι όντως είναι μία από τις τρεις ε, αυτές οι καταγγελίες, η καταγγελία ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Συνδικάτου, αλλά με δεσμεύουν οι κανόνες της ε, εμπιστευτικότητας του απορρίτου. Επιβεβαιώνω λοιπόν ότι έχουμε λάβει υπόψη την καταγγελία αυτή. Πρόκειται για μία παρέκκληση πρώτου τύπου, όπου ο έμεσος εργαζόμενος ε, έχει μόνιμο συμβόλαιο και πληρώνεται μεταξύ των συμβάσεων έργου. Και αυτό έχει να κάνει με τη διαφορά μισθού που έχει ο έμεσος εργαζόμενος σε σχέση με το επίπεδο μισθού που έχουν οι κανονικοί εργαζόμενοι. Έχουμε έρθει σε επαφή με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τις πιλωτικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε θέσει και κάποια σημεία επαφής με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγκρεμεί η υπόθεση και έχετε δίκιο. Έχει έρθει η ώρα να αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα κλείσει την υπόθεση ή θα προχωρήσει σε διαδικασία επί παραβάση. Και ελπίζω να το κάνει σύντομα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα όμως δεν έχουμε χρονοτριβήσει σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Συλλέγουμε πληροφορίες και από τον καταγγελων, από τον καταγγέλλοντα και από τις εθνικές αρχές και πλέον έχουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να λάβουμε μια απόφαση. Αλλά πολύ φοβάμαι δεν μπορώ να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Ο κύριο Σάιμον, για να δευτερολογήσει. Σας ευχαριστώ. Να διευκρινίσω το εξή. Είναι περίεργη αυτή η ιδέα ότι δεσμεύεστε από την αρχή τη Εμπιστευτικότητα. Μιλάμε για την Επιτροπή απασχόληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια, ένα σώμα που έχει εκλεχθεί ακριβώ για να ελέγχει αυτά που κάνετε. Πρόκειται για μια δημόσια καταγγελία. Έχω ανακοινωθέν τύπου του TUC, του συνδικάτου, TUC, του, της τρίτης... Ε, της Συνομοσπονδία Συνδικάτων TUC τη 3η Σεπτεμβρίου 2013. Πείτε μας λοιπόν, τι σας δεσμεύει για εμπιστευτικότητα. Και μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτό που μάλλον λέτε, ότι παρά την ρήτρα εμπιστευτικότητας, σκοπεύετε να απαντήσετε σύντομα στην καταγγελία της Συνομοσπονδίας μετά από 15 μήνες. Είπατε τώρα ότι τώρα έχει έρθει ο χρόνος να απαντήσετε. Μπορούμε να περιμένουμε απάντηση πριν τα Χριστούγεννα. Η απάντηση. Όταν γίνεται μια καταγγελία, ο καταγγέλων έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητα. Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι δεν το κάνουν. Στην προκειμένη περίπτωση η Συνομοσπονδία ζήτησε εμπιστευτικότητα. Το τι έκανε στη συνέχεια με τα ανακοινωθέντα τύπου δεν μας αφορά. Εμάς μας δεσμεύει η ρήτρα εμπιστευτικότητας όταν το ζητάει ρητά ο καταγγέλων. Σχόλιο εκτός μικροφώνου από τον κύριο Σάιμον. Under what Υπό ποιο καθεστώ έρχεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας λέτε ότι είναι εμπιστευτικές οι πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να μου αποστείλετε επακριβώς ε, και γράφος της ε, το καθεστώς αυτό. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Να σας πω ότι όπως σας ανέφερα, έχουμε, είχαμε επαφές και με τον καταγγέλλοντα, συναντηθήκαμε και με τις εθνικές αρχές σε διάφορες περιστάσεις, εκρεμεί ακόμα η υπόθεση, είναι ανοιχτή η υπόθεση. Και η απόφαση θα ληφθεί από την πολιτική αρχή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν τυχόν αποφασιστεί ε, διαδικασία επί παραβάση. Κυρία Στάινρουκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο και δεν μας ικανοποιεί καθόλου όταν διαρκεί τόσο πολύ η εφαρμογή και παραμένουν εκκρεμή τόσα πολλά ζητήματα σε ό,τι αφορά τις μισθολογικές ε, αμοιβέ, τις ε, διακοπές. Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο θα αντικαταστήσει το μόνιμο προσωπικό από πιο ε, ελαφριές συνθήκες εργοδοσίας. Ήμουν ε, επί πέντε χρόνια ε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης για την Εύρεση Εργασίας στην περιφερειά μου και ήδη τότε διαπιστώσαμε, διαπιστώναμε ότι δεν πρόκειται για μια γέφυρα προς μια πιο μόνιμη μορφή εργασίας, αλλά μάλλον ένα διέξοδο. η επάνωδο στην κανονική αγορά εργασία είναι κάτι το σπάνιο και μάλλον καταλήγουν σε μια μόνιμη επισφαλή απασχόληση τα άτομα αυτά. Μπορείτε να αξιολογήσετε, γιατί τα δεδομένα τα έχετε μάλλον στη διάθεσή σας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Από ό,τι μας λέτε, είναι μη ικανοποιητική. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν υπάρχει ανάγκη βελτίωσης, μας λέτε. Για εξηγήστε μας, σε ό,τι αφορά την ερμηνεία του άρθρου 4, περιμέναμε απόφαση από τον Οκτώβριο. Χαίρομαι λοιπόν που την περιμέναμε τώρα την απόφαση. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχουν κίνδυνοι να υπάρχει περισσότερη αντικατάσταση κανονικών μορφών εργασίας από τις έμεσες αυτές μορφές απασχόλησης. Δηλαδή μια αρνητική διαμόρφωση της κατάστασης για τους εργαζόμενους. Έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα σε θέματα εφαρμογής. Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα δηλώνουν ότι για παράδειγμα στη Γαλλία, στο δημόσιο τομέα, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αντικατασταθούν από τέτοιου έμεσου εργαζόμενου. Γνωρίζετε την κατάσταση στη Γερμανία. Πολύ καλά. Δεν τηρείται η αρχή τη ίση μεταχείρισης. Το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου το έθιξε άλλωστε και συνάδελφο ήδη. Και διαβουλευσει με τους κοινωνικού εταίρου σε κάποια κρατημέλη δεν κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση, στη Βουλγαρία για παράδειγμα ή στην Πορτογαλία. Μπορείτε να σχολιάσετε και τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ το συντομότερο δυνατόν σε δύο χρόνια το αργότερα να έχουμε μία έκθεση εφαρμογής η οποία και να δημοσιευθεί. Γιατί μπορούν να ανακύψουν προβλήματα σε πάρα πολλούς τομείς. Και είπα τα τελευταία ερώτηση ότι σε κράτη-μέλη έγιναν ε, έρευνες και ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τα προβλήματα. Ρωτήσατε που είναι τα προβλήματα για τους εργαζό... εργαζόμενους και για τους μόνιμους κανονικούς εργαζόμενους και για τους έμεσους επασχολέμενους. Γιατί στατιστικά αν αυξάνεται η έμεση, η έμεσα απασχολούμενη, μειώνονται οι κανονικά απασχολούμενοι. avec la consultation Um, um, uh, Πρέπει να πω ότι ο σκοπός της οδηγίας δεν είναι να περιορίσει τη χρήση των προσωρινά εργαζόμενων. Αντιθέτως, σκοπός της οδηγίας είναι να αναγνωρίσει, να νομιμοποιήσει το, της, ε, την απασχόληση μας προς προσωρινή απασχόλησης; Με την αρχή της ίσης απασχόλησης. Στο βαθμό λοιπόν που οι όροι εργασία των προσωρινά εργαζόμενων βελτιώνονται λόγω της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει εμπόδιο για την περαιτέρω χρήση τέτοιου τύπου εργασίας. Αυτή είναι η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από την οδηγία. Μα μας ικανοποιεί στο 100% η εφαρμογή. Όχι, σας το είπα. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πολύ στενά την εφαρμογή της οδηγίας. Ως τώρα όμως δεν έχουμε δει συγκεκριμένη πρόταση τροποποίηση της οδηγίας και καμία επιθυμία δεν έχει εκφραστεί ούτε από τα κράτη-μέλη ούτε από τους εμπλεκόμενου φορείς να τροποποιηθεί η οδηγία. Θεωρούμε ότι η εργασία μέσω προσωρινής απασχόλησης έχει την χρήση της ιδιαίτερα σε περιστάσεις όπου δεν υπάρχει σαφές ε, οικονομικό μέλλον, όπου δεν ξέρουν οι επιχειρήσεις για πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστούν να απασχολήσουν κάποιους εργαζόμενους. Υπάρχει κάποια μορφή προκειμένου με τον τρόπο αυτό. Μπορεί να είναι δραστηριότητε εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονε σε, σε μικρόμεσες επιχειρήσεις δεν έχουν τις δυνατότητε και τους πόρου να κάνουν τι απαραίτητε έρευνε και μελέτε. Άρα χρησιμοποιούμε έτσι τους καλύτερους τρόπους. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει αρνητικό αντίκτυπος. Θεωρούμε ότι αυτοί οι προσωρινά εργαζόμενοι λαμβάνουν έτσι τις σωστές ε, συνθήκες εργασίας, την κατάλληλη προστασία σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την προστασία, την, προστα... την πρόσβαση σε άλλες ε, υπηρεσίες. Το θέμα είναι σε τι βαθμό παραβιάζονται οι αρχές αυτές. Δεν θέλουμε η αρχή της συμμεταχείρισης να είναι θεωρητική αρχή και να μην αφορά την πράξη. Κοιτάμε, για παράδειγμα, την παρέκκληση της Σουηδίας και της, του Ηνωμένου Βασιλείου, να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα, ποια είναι οι διαφορές, ποια είναι τα διαφορετικά αποτελέσματα στα οποία μπορεί να οδηγήσει η παρέκκληση. Άρα, υπάρχει δυναμικό βελτίωση, βελτίωσης, ναι. Σας ανακοίνωσα ποια είναι τα εργαλεία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχά, διαδικασία επί παραβάση. Όταν θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν επαρκώς την οδηγία. Κατά δεύτερο, συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ναι, ζητήσαμε και τη γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων σε ό,τι αφορά την λειτουργία τη οδηγία λάβουμε καταγγελίες από τα συνδικάτα σε ό,τι αφορά κάποιες πτυχέ τη εφαρμογή τη οδηγία. Ωστόσο, δεν ε, ζητήθηκε τροποποίηση τη οδηγία από τα συνδικάτα. Αυτά, λοιπόν, είχα να σας αναφέρω. Τώρα, και πάλι το θέμα της μεταβατικής ε, φάσης. Τα πλαίσια της μελέτης αυτής δεν κάναμε αξιολόγηση, ε, δεν κάναμε σε ό,τι αφορά το ποσοστό των ατόμων για τα οποία η φάση της προσωρινής απασχόλησης αποτελεί μια μεταβατική φάση προς τη μόνιμη απασχόληση. Υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει από κάποιες εταιρείες συμβουλευτικής από τον ίδιο τον οικονομικό κλάδο που μας έχουν χορηγήσει κάποια αριθμητικά στοιχεία. Αλλά στα πλαίσια της έρευνας αυτής, της προκειμένης, δεν έγινε τέτοια έρευνα. Thank you. I'll give the floor. Σας ευχαριστώ. κυρία κάνει και την ερώτηση για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα κράτη-μέλη. Μπορείτε να μας πείτε αν ισχύει ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή της οδηγίας δεν συμπεριλήφθησαν οι κοινωνικοί εταίροι και τι έκανε η Κομισιόν σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι κάτι που είναι στην οδηγία. Ε? the implication Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων γίνεται σε διάφορα επίπεδα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι, συμμετέχουν στην ομάδα εμπειρογνωμόνων και συμμετείχαν πλήρω και στην εκπόνηση της έκθεσης. Στα κράτη-μέλη ε, προβλέπεται εξάλλου διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για την υποβολή των εθνικών εκθέσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι, εάν τελικά δεν έχουν αυτό το δικαίωμα να αποφανθούν με τη μέσω διαβούλευση σε επίπεδο κράτους μέλους μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο Απαιτείται η συμμετοχή ε, των κοινωνικών εταίρων μέσα από διαδικασίες ε, σύναψης συλλογικών ε, συμβάσεων. Είναι ένα θέμα που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή και αποκλήσεις για την ίση αμοιβή δεχόμαστε μόνο όταν εφαρμόζεται σωστά η συλλογική σύμβαση εργασίας. Και αυτό το θέμα το μελετούμε τώρα. Αυτά έχω να σας πω προς το παρόν. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα δύο ερωτήσεις, ε, μάλλον δύο ομιλητές. Κύριος Ούλη Κρίστενσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον ε, κύριο Σίλβα. Νομίζω το Δεκέμβρη του 2009 ήταν που συμφωνήσαμε αυτήν την οδηγία. Ε, ε, συμφωνήσαμε για την ε, έγκριση αυτής της οδηγίας. Ήταν μεγάλη σημαντική μέρα για το Κοινοβούλιο γιατί δεν υπάρχουν και πολλά νομοθετήματα σε αυτό το τομέα. Εγώ είμαι υπέρ της αυξημένης ευελιξίας στην αγορά εργασίας ούτως ώστε να εισέλθουν περισσότεροι ε, εργαζόμενοι και μετά από μία μεταβατική περίοδο να περάσουν σε μόνιμες θέσεις απασχόλησης. Το πρόβλημα όμως είναι ότι με όλες αυτές τις εξαιρέσεις δεν είναι ποιοτική η παρέμβασή μας και δεν δημιουργούνται οι λύσεις που χρειαζόμαστε. Ο στόχος των εξαιρέσεων τελικά είναι η αποφυγή της ίσης αμοιβή και έτσι καταρρύπτεται το βασικότερο επιχείρημα για την εφαρμογή μιας τέτοιας νομοθεσίας. Ε, δηλαδή προσπαθούν όλοι να βρουν τρόπους παράκαμψης του νομοθετήματος. Εμείς επιθυμούμε να εφαρμοστούν θεμητοί όροι ανταγωνισμού, όπως ήταν και ο στόχος της οδηγίας, δηλαδή να είναι ισότιμη μεταχείριση για τους προσωρινά απασχολούμενους, να ε, είναι θεμητοί όροι ανταγωνισμού και για τους προσωρινά ε, απασχολούμενος και για τους μόνιμα απασχολούμενους. Ε, δεν θέλουμε να σκοτώνονται μεταξύ τους οι εργαζόμενοι. Υπάρχει κάποια εγγύηση που μπορείτε να μας δώσετε. Ευχαριστώ κύριο Μάν. Okay. Ευχαριστώ. Αυτό το θέμα της εμπιστευτικότητας το έλεξα. Ε, σωστό είναι αυτό. Αλλά θέλουμε ως Επιτροπή να μάθουμε τι έχει γίνει θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια οδηγία για να βγουν από αυτή την κρίζα ζώνη όλες αυτές οι εταιρείες ΕΠΑ να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Στη Γερμανία επισκέφθηκα μερικές τέτοιες εταιρείες και εξεπλάγει για το πόσες ρυθμίσεις έχουν ήδη εφαρμόσει με σωστό τρόπο. Όμως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την κατάσταση με την κατάσταση σε διάφορες τέτοιες εταιρείε σε άλλες χώρες. Γι' αυτό ρωτάω. Μας είπατε ότι έχετε μόνιμη ανταλλαγή απόψεων με τους κοινωνικούς εταίρους. Και ορισμένες από τις απαντήσεις τους τις λαμβάνουμε και εμείς. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η επιτροπή που έχετε δημιουργήσει είναι επαρκής για να μπορεί να συλλέξει πληροφόρηση ηλεκτρονικός. Βεβαίως γίνεται, αλλά πρέπει να συνεδριάζει σχετικά συχνά. Και δεύτερον, εμείς στο Κοινοβούλιο είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος των κοινωνικών εταίρων, αλλά ξέρω ότι πολλοί κοινωνικοί εταίροι δεν είναι στο επίπεδο λειτουργίας, δεν υπάρχουν όπως θα θέλαμε. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε να δημιουργηθούν τέτοιοι κοινωνικοί εταίροι. Και στις, ε, στα πορίσματα είπατε ότι θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε και το ευρωπαϊκό εξάμεινο, δηλαδή να κάνετε συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα δεν είναι ήδη θεσμοθετημένο αυτό. Ακόμη πρέπει να εφαρμοστεί και όπως είπε και ο Όλεϊ, Αναφερθήκατε στην ευελιξία στην αγορά εργασία. Είπαμε ναι ότι πρέπει να είναι ευέλικτη αλλά και ασφαλή η απασχόληση. Αλλά είπατε ότι ο ρόλος της προσωρινής εργασίας πρέπει να ε, προσαρμοστεί στις ε, συνθήκες ε, της σύγχρονης εργασίας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της κυρίας Στάιμπρουκ, ότι μπορεί να οδηγήσει σε επισφάλεια. Μπορείτε να μας δώσετε τη δική σας άποψη για το τι σημαίνει ευελιξία στην σύγχρονη εργασία. Ο κύριος Σίλβα, παρακαλώ. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, μας πήρε έξι χρόνια για να εγκριθεί η οδηγία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες συζητήσεις που έγιναν στο Συμβούλιο. Περιστρέφονταν κυρίως γύρω από το θέμα των εξαιρέσεων. Σε ορισμένες χώρες όπου υπάρχουν λιγοστέοι περιορισμοί για την χρήση των εταιριών προσωρινής απασχόλησης, δεν μπορούσε να γίνει εύκολα δεκτή εισαγωγή ρυθμίσεων για την ίση αμοιβή, Φερπίν. Και επειδή υπάρχει αυτή η περίοδος δοκιμής, ε, ε, και αυτό μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Ε, χρειαστήκαμε έξι χρόνια γιατί είναι πάρα πολύ διαφορετικές οι εθνικές ρυθμίσεις για αυτήν την περίοδο. Και ξαναλέω, τα κράτη-μέλη δεν ζητούν αυτή τη στιγμή αναθεώρηση της οδηγίας. Δεδομένου του αριθμού των καταγγελιών που έχουν λάβει θεωρούν ότι δεν δικαιολογείται η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Σίγουρα υπάρχουν άλλες οδηγίες στον τομέα αυτό που χρήζουν αναθεώρησης. Πάλι επί τη βάση των καταγγελιών ε, που λαμβάνουμε των διαδικασιών επί παραβάση που βασίζονται σε αυτές τις καταγγελίες δεν κρίνουμε εμείς ότι συνιστά προτεραιότητα η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Θέλω να είμαι σαφής γι' αυτό. Ναι, θέλουμε να ε, ρυθμίσουμε τα προβλήματα διότι υπάρχουν και εντοπίστηκαν στην εφαρμογή της οδηγίας σε πώς χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη παραδείγματος χάρη το άρθρο 4 για την αναθεώρηση των εξαιρέσεων αλλά και για την εφαρμογή κάποιων εξαιρέσεων οδηγεί σε καταστάσεις που πόρο απέχουν από ισότιμη μεταχείριση. Αυτά τα προβλήματα προσπαθούμε να ρυθμίσουμε, στα πλαίσια όμως την οδηγία πάντως δεν έχουμε καμία πρόθεση να την αναθεωρήσουμε. Δεν τίθεται το ζήτημα. Η ευελιξία που προσφέρει η οδηγία συνίσταται στη χρήση άνευ περιορισμών της προσωρινής απασχόλησης, όπως ε, η κλαδική απαγόρευση ή ο χρονικός περιορισμός ε, των συμβάσεων σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το βασικό παράπονο των επιχειρήσεων, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προσωρινή απασχόληση στο μέτρο που θα ήθελαν λόγω των ενισχύ εθνικών περιορισμών. Τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτό. Η οδηγία ε, δράζεται επί το άρθρο 153 το άρθρο 153 της Συνθήκης προσδίδει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση την αρμοδιότητα να νομοθετεί για να προστατεύσει μέσω ελαχίστων προτύπων τους εργαζομένους. Οι επιχειρήσεις θέτουν αυτό το ζήτημα το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί στα πλαίσια ενός άλλου νομοθετήματος ε, που αποσκοπεί στην θέσπιση εργαλείων εναρμόνισης ε, για ελεύθερη πρόσβαση στις ΕΠΑ. Αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια νομοθεσίας για την ενιαία αγορά και όχι για το εργατικό δίκαιο. Μπορούμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν τους περιορισμούς, όμως σε καμία περίπτωση οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να ζητήσουν να επιβάλλουμε εμείς την άρση των εθνικών περιορισμών. Δεν έχουμε νομική βάση, δηλαδή, μέσα σε αυτή την οδηγία για να επιβάλλουμε την άρση των περιορισμών. Συστήνουμε ευελιξία, συστήνουμε να επιβάλλονται αναλογικοί περιορισμοί. Μόνο συστάσεις μπορούμε να κάνουμε, όμως τίποτα παραπάνω. Για την προστασία των εργαζομένων, όπως έλεγα, Εξετάζουμε τις αναφορές, τις καταγγελίες και τα αιτήματα για διαδικασία επιπαραβάση από τους πολίτες. Ε, είμαστε σε διαρκή επαφή με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για αυτά τα ζητήματα. Και όπως σας είπα, Αυτό που προσπαθούμε είναι να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν οδηγία με τρόπο που να συνάδει με τους στόχους της. Ευχαριστούμε. Αγκύρ και Μαρτά. Grazie Presidente, eh, vorrei partire da, da una considerazione. Innanzitutto che... Θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο. οι συμβάσεις αυτές όταν μιλάμε για συμβάσεις περιορισμένης διαρκείας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται με τις εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις και αυτές θα πρέπει να προστατεύονται. Κάτι άλλο να υπογραμμίσω σε ό,τι αφορά την κινητικότητα στην αγορά της εργασίας. Μιλάμε πάντα για την αρχή αυτή της κινητικότητας, αλλά θεωρώ ότι πρόκειται για μια επισφαλή μορφή εργασίας, όπου δεν υπάρχει εγγύηση της κοινωνικής προστασίας. Σε ό,τι αφορά τις, ε, την σωστή εφαρμογή των εργασιακών συνθήκων για να υπάρχει μια σωστή προστασία. Αυτό ήθελα να το πω εξ αρχής. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, ρυθμίσεις ε, κατεξαίρεση. Χρησιμοποιείται αυτό πάντα ως δικαιολογία για να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι τους αρέσουν. Και με, το, ε, με τις ρυθμίσεις της εξαιρετικών περιστάσεων υπάρχει αυτή η δικαιολογία λοιπόν για να κάνουν ό,τι θέλουν. Σε κάποια φάση λοιπόν υπήρχε η γερμανική παρέκκληση, υπάρχουν άλλες παρεκκλήσεις. Οι παρεκκλήσεις έχουν να κάνουν με την αμοιβή μόνο. Ή γενικότερα σε ό,τι αφορά τις γενικότερες ρυθμίσεις. Γιατί φυσικά και το μισθό, οι αποδοχέ θα πρέπει να είναι οι ίδιε, αλλά και οι όροι εργασία. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Μαρτά. Ευχαριστώ. Με βάση την συζήτηση που έχει γίνει, διαπιστώνουμε ότι η χρήση αυτής της μορφής εργασίας ε, ποικίλει πολύ από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένες χώρες τελικά είναι εκμετάλλευση. Δεν υπάρχει συμμεταχείριση, δεν υπάρχει ασφάλεια, τίποτα. Στη Γαλλία συνολικά είναι πολύ καλή η κατάσταση. Είναι καλή η χρήση αυτή τη μορφή εργασία και οι επιχειρήσει είναι πολύ ικανοποιημένε. Ερωτήσει. Πρόκειται να ορίσετε ε, ε, μέγιστο ποσοστό απασχολουμένων τέτοιου τύπου για να αποφευχθούν κατά χρήση, δηλαδή 80% να είναι προσωρινά εργαζόμενοι. Αυτό θα ήταν κατάχρηση. Και επιπλέον σκοπεύουμε να περιορίσουμε την εκτέλεση των ίδιων καθηκόντων επανειλημμένα μέσω προσωρινής απασχόλησης γιατί αυτό θα σημαίνει ότι τελικά ποτέ δεν πρόκειται να προσλάβει μόνιμο κάποια εταιρεία. Επίσης έχουμε και ειδικού της προσωρινής εργασίας εδώ είναι οι διερμηνείς μας και εποφελούμε να τους συγχαρώ για τα θαυμάσια εργασία τους. Λοιπόν, για την πρώτη σας ερώτηση της ε, Ιταλίδας ε, ε, ε εάν δεν είχαν υπάρξει εξαιρέσεις δεν υπήρχε υπάρξει οδηγία να είμαι σαφής αυτή ήταν η κατάσταση το 2008 χωρίς εξαιρέσεις δεν είχαμε καταλήξει οδηγία δεν είναι λοιπόν ρεαλιστικό να θεωρήσουμε ότι θα έχουμε μια οδηγία που θα καθορίζει προδιαγραφέ προστασία των εργαζομένων χωρί εξαιρέσει. Είναι η μόνη δυνατότητα εξαιρέσει να έχουμε κάποιου ελάχιστου κανόνε που εφαρμόζονται σε 28 κράτη-μέλη με τόσο διαφορετικές καταστάσεις από πλευράς ε, θεσμών, κανόνων και περιορισμών για την προσωρινή εργασία. Είναι ελάχιστες οι προδιαγραφές αυτές αν το επιθυμούν. Τα κράτη-μέλη μπορούν να επιβάλλουν θετικότερα επίπεδα προστασίας. Αυτά είναι, αυτές είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που ε, μπορέσαμε να επιτύχουμε. Χωρίς εξαιρέσεις δεν θα υπήρχε οδηγία για την ερώτηση που θέσατε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει να επιβάλλει ποσοστώσεις για την προσωρινή απασχόληση στις επιχειρήσεις. Αυτό θεωρώ ότι θα ήταν ε, μικροδιαχείριση. Αυτό νομίζω ότι θα παραβίαζε κάθε λογική επικουρικότητας. Όχι. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Προσπαθούμε να εγγυηθούμε την ίση μεταχείριση στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο του δυνατού την προστασία των προσωρινά εργαζομένων. Όχι, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τέτοιου τύπου περιορισμούς στις επιχειρήσεις. Τώρα για την ερώτηση για τις καταχρήσεις, δηλαδή ότι επανειλημμένα κάποια συμβόλαια για το ίδιο καθήκον να είναι προσωρινής εργασίας. Στο βαθμό που ε, ένα μεγάλο τμήμα των προσωρινών εργαζομένων έχουν ε, συμβόλαιο ορισμένου χρόνου προστατεύονται από τον υπερβολικό αριθμό διαδοχικών ε, συμβολέων από την οδηγία που ρυθμίζει την ε, εφαρμογή των συμβολέων ορισμένου χρόνου. Είναι η 99 κάθετος 2011. Υπάρχει αυτή η οδηγία που καθορίζει τον μέγιστο αριθμό συμβολέων ορισμένου χρόνου. Και αν είναι προσωρινά εργαζόμενοι, αυτομάτω υπάγονται σε αυτή την οδηγία. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα των προσωρινών εργαζομένων που έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι έχουν εργασία προστατευόμενη, αλλά μετατίθενται από διάφορες επιχειρήσεις από μία επιχείρηση σε άλλη και εκεί δεν υπάρχει περιορισμός. Αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι η κύρια εργασιακή σχέση με τον εργοδότη τους, η οποία ε, υπάγεται σε συμβόλαιο αορίστου χρόνου. Σας ευχαριστώ. Τώρα το ερώτημα του κυρίου Σούλτς και μετά τον κύριο Φουντούλη. Ε, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και τις εξηγήσεις σας. Έχω μία ερώτηση και μία παρατηρήση να κάνω. Καταρχάς, η ερώτηση. Έχετε εμπειρίες σε ό,τι αφορά την σχέση μεταξύ της ε, προσωρινής απασχόλησης και του κατώτατου μισθού. Σε κάποιες χώρες ε, υπάρχουν κατώτατοι μισθοί, κάποιες άλλες εισήγαγαν κατώτατο μισθό τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει επιρροή από τις θέσεις προσωρινής απασχόλησης. Τώρα, για την παρατήρησή μας, ε, την παρατήρησή μου, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το καθεστώς προσωρινής απασχόλησης μπορούμε να ενημερωθούμε μέσω μελετών κτλ. Αλλά αυτό που με εντυπωσιάζει όταν ε, ξεκινάω εδώ στο κοινοβούλιο μετά από 10 χρόνια στις επιχειρήσεις είναι ότι διαπιστώνω ότι όταν ε, δεν μεταχειριζόμαστε με σωστό τρόπο τους προσωρινά απασχολούμενους δεν είναι αντίστοιχα και τα αποτελέσματα. Μάλλον είναι αντίστοιχα και τα αποτελέσματα. Είναι χαμηλότερα τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η εμπειρία μου από τη Γερμανία. Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Στάινρουκ δεν μπορώ να πω ότι με βρίσκουν σύμφωνο. Και αυτό λέει η εμπειρία μου, η δεκαετής εμπειρία μου, ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από την πλευρά μας, γιατί με την εφαρμογή της οδηγίας αυτής εξυπηρετούνται, μήπως μάλλον με την εφαρμογή της οδηγίας αυτής, εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των μεγάλων εργοδοτών, έτσι ώστε να έχουν εργαζόμενους με χαμηλό, κόστο, χωρί κόστος, δικαιώματα, γιατί είναι γνωστό ότι με τη μέθοδο της εργασίας μέσω, μέσω εταιριών προσωρινής απασχόλησης σε πολλές χώρες καταστρατηγούνται τα εργασιακά δικαιώματα. Έχω ιδιαίτερη αντίληψη από τη χρήση ενοικιαζομένων εργα... ας μου επιτραπεί η έκφραση ενοικιαζομένων εργαζομένων στα ελληνικά ταχυδρομεία, όπου η εταιρεία χρησιμοποιεί τους εργαζόμενους κατά το δοκούν, δύο ώρες το πρωί, δύο ώρες το απόγευμα, ανάλογα με την κρίση του έμεσου εργοδότη, αδιαφορώντα όμως για τις επιπτώσεις στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή τους. Η οδηγία θα έπρεπε να επανεξεταστεί στο σύνολό τη. Συζητάμε για ισότιμη μεταχείριση μεταξύ ποιών, μεταξύ των μονίμω απασχολουμένων και των ορομιστίων, να το πω έτσι. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι θέσει εργασία με μόνιμη απασχόληση. Η οδηγία προφανώ, ίσω χωρί να το ξέρουμε, θέλει να ονομιμοποιήσει τι εταιρείε που εκμεταλλεύονται την ανάγκη για εργασία των πολιτών και εισπράττουν χρήματα μεσητείας ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους εργοδότες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σίλβα για να απαντήσει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει μελέτη πριν από κάποια χρόνια για την ε, επισφαλή φύση των θέσεων εργασίας. Και ναι, διαπιστώσαμε λοιπόν ότι υπάρχουν τέτοιες ε, επισφαλείς συνθήκες. Δεν αρνούμε ότι υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις και αυτές οι περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι χωρίς την οδηγία αυτή θα ήμασταν σε χειρότερη θέση. Αυτή η οδηγία έχει θέσει κάποιους όρους προστασίας για την προστασία των εργαζομένων που δεν υπήρχαν πριν σε κάποια από τα κρατη Χωρίς την οδηγία δεν θα υπήρχαν κανόνες προστασίας για τους εργαζόμενους αυτούς που αποτελούν το 1,6% του εργατικού δυναμικού και σε κάποιες χώρες ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Κάποια κράτη-μέλη αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν στην εθνική τους νομοθεσία και κανόνες που είναι πιο υψηλής προστασίας από αυτό που υπήρχε προηγουμένως. Άρα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατευθύνση σε ό,τι αφορά την προστασία των εργαζομένων για τους κατώτατους μισθούς. Ναι, ναι, φυσικά και ισχύει. Για τους προσωρινά απασχολούμενους, με ή χωρίς οδηγία. Αλλά η προστασία που επιθυμούμε εδώ είναι πάνω από το επίπεδο του κατώτατου μισθού. Γιατί μιλάμε για ίση μεταχείριση με τους εργαζόμενους που κάνουν αντίστοιχη δουλειά στην ίδια εταιρεία. Άρα το θέμα του κατώτατου μισθού δεν είναι ιδιαίτερα σχετικό εδώ. Προσπαθούμε να περάσουν όροι και συνθήκες πάνω, πολύ πιο πάνω από το κατώτατο μισθό. Ε, πρόκειται για ένα ελάχιστο επίπεδο αποδοχής, αποδοχών. Η κυρία Μάκιντάιρ και η κυρία Μορβάη στη συνέχεια. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σίλβα, για την παρουσίασή σας. Πολύ ενδιαφέρουσα τη βρήκα. Και εγώ είμαι από το χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 25 χρόνια είχα επιχείρηση, όπως και άλλοι που μίλησαν νωρίτερα. Ε, δεν θα τα καταφέρναμε, πρέπει να σας πω, αν δεν χωρίς τους προσωρινά αποσχολούμενους Δηλαδή, όταν κάποιο παίρνει την αιτήσια άδεια, τι κάνετε. Παίρνετε ένα προσωρινό αποσχολούμενο να έρθει να καλύψει το κενό. Ή κάποιο αρρωστήσει, παραδείγματο χάρη. Πρέπει να έχετε τη δυνατότητα αυτή. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απασχόληση. Δηλαδή, μπορεί κάποιον να τον έχετε απασχολήσει προσωρινά, του έχετε συνηθίσει, του ξέρετε, σα ξέρουν. Εάν ε, ανακύψει μία ανάγκη, τότε είναι η φυσιολογική επιλογή. Δεν θέλω να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι είναι κακή η προσωρινή ή και η μερική απασχόληση. Οι τι θέλουν την μερική απασχόληση. Ας μην φύγουμε από τη σημερινή συνεδρίαση πιστεύοντας ότι είναι κακό πράγμα η προσωρινή απασχόληση και επιτρέπεται μόνο ε, υπό ορισμένε συνθήκε. Δεν μπορεί να επιβιώσει καμία επιχείρηση. Και δεν μιλάω μόνο για την ετήσια άδεια, την αναρωτική και τα κενά που καλύπτονται. Έχετε ένα σχέδιο και θα σα πάρει κάποιου μήνε να το ολοκληρώσετε. Τι θα κάνετε, θα προσλάβετε και μετά θα έχετε υπεράριθμο προσωπικό. Όχι, θα προσλάβετε κάποιον προσωρινά και θα διαχειριστεί μέχρι την περάτωση του έργου αυτό το ε, πρόγραμμα. Και θέλω να ακουστεί και η άλλη πλευρά. Ε, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η δυνατότητα προσωρινή απασχόλησης. Λοιπόν, για να κάνω και τις ερωτήσεις μου. Τρεις καταγγελίες είναι ελάχιστο αριθμό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι κατάλαβα. Και ο Τζον Σάιμον μας είπε ότι η μία καταγγελία ήταν από τα Βρετανικά Συνδικάτα. Εγώ αναρωτιέμαι, Έχετε λάβει καταγγελίες σε σχέση με το άρθρο 4 περί τι περιορισμοί ή απαγορεύσεις, αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου, έχετε λάβει σχετικές καταγγελίες. Ευχαριστούμε κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Μακιντέιρ ευχαριστω κυρια προεδρε η κυρια μακιντειρε ζητησε το λόγο και εγώ γέλασα λίγο. Καλύτερα να είχα κλάψει όμως. Γιατί Εδώ καταδεικνύεται εκ νέου ότι ζούμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Τα παλιά κρατημέλη και τα καινούργια, τα απεικιοκρατημένα κρατημέλη, στα οποία συγκαταλέγεται και η πατρίδα μου. Για την Ουγγαρία το φαινόμενο αυτό, η προσωρινή απασχόληση, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ε, ανέφερε η κυρία Μάκιντάιρ. Να σας πω λοιπόν και να σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους στην Ουγγαρία. Ότι οι δυτικέ εταιρείε οι οποίες παραγούν στην Ουγγαρία απασχολούν μόνο προσωρινούς επασχολούμενους και εργαζόμενους. Δεν έχουν κανονικό προσωπικό, μόνιμους υπαλλήλους. Γιατί? για να στερήσουν όσο πιο πολλά δικαιώματα γίνεται από τους εργαζόμενους. Και με 200-300 ευρώ είναι μοντέρνη σκλάβη ουσιαστικά. Αυτό σημαίνει για μας ε, αυτό το φαινόμενο. Ακόμα και αυτό το, αυτός ο όρος ε, της δανειζόμενης εργασίας. Ε, δανείζουμε σκούπες ηλεκτρικές, δανείζουμε DVD, όχι ανθρώπους. Στην Ουγγρική λοιπόν, ε, στους, με ουγγρικούς όρους μιλάμε για δανειζόμενους εργαζομένους. Υπάρχουν ε, επιχειρήσεις που δανείζουν και επιχειρήσεις που δανείζονται. Μιλάμε για ανθρώπους. Πού είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και έχω λοιπόν μια συγκεκριμένη ερώτηση να σας κάνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρει πως ε, γίνεται κατάχρηση των δυνατοτήτων αυτών. Και σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που εκπροσωπούνται σε αυτή την ad hoc επιτροπή, ποιος εκπροσωπεί τους Ούγγρους εργαζόμενους, έχετε μια συγκεκριμένη απάντηση να μου δώσετε. Και άλλη μια ερώτηση, ξέρετε με τι άσχημες ε, συνθήκες εργάζονται οι Ούγγροι εργαζόμενοι για τις δυτικές εταιρείε. Τα ξέρετε αυτά. Και ξέρετε ποιες είναι οι εμπειρίες των Ούγγρων εργαζομένων. Um, uh, λοιπόν, να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας ε, Μακιντάρ. Ναι, μία από τις ενστάσεις υποβλήθηκε από μια οργάνωση εργοδοτών της Σουηδίας και αφορά το άρθρο 4 το θέμα των περιορισμών και το πώς η κυβέρνηση, η συγγνώμη, η σουηδική κυβέρνηση διαχειρίζεται αυτούς τους περιορισμούς και η τρίτη ένσταση είναι από ένα γερμανό πολίτη και αφορά τη διάρκεια των ε, ε, χορηγιών εργαζομένων σε εταιρείες πρέπει να πω ότι η Επιτροπή επίσης έλαβε θέση έναντι του κράτους μέλους που δεν υπέβαλε έκθεση για την εξέταση των ε, περιορισμών. Η χώρα αυτή όπως αναφέρεται στην έκθεση είναι το Λουξεμβούργο, είμαστε σε επαφή με τις αρχές του Λουξεμβούργου για να μας απαντήσουν. Για τις συνθήκες εργασίας στην Ουγγαρία, τα ουγγρικά συνδικάτα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά συνδικάτα, στις ευρωπαϊκές συνομοσπονδίες συνδικάτων, έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους και να πούν στην ομάδα εμπειρογνωμόνων ποια είναι τα προβλήματα σε αυτήν την επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και υπάρχει επίσης και μια ειδική κλαδική επιτροπή ιδιαίτερα για τα θέματα των ε, εργαζομένων μέσω εταιριών προσωρινής απασχόλησης. Και επίσης έχουμε εκπροσώπους των εργαζομένων από όλες τις χώρες της Ευρώπης, εκπροσώπους των εργαζομένων της προσωρινής απασχόλησης και αυτά τα θέματα ανακύπτουν σε αυτόν τον ε, διάλογο, ε, τον κλαδικό για τα κοινωνικά θέματα. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Σίγουρα θα έχουμε δυνατότητα να επανέλθουμε αργότερα. Το 7, το 7 Με συγχωρείτε να συνεχιστεί η συζήτηση εκτός της ε, αίθουσας. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013. Ο κύριος Κάζα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για τις τροπολογίες που υποβάλλατε στη γνωμοδότησή μου. 88 τον αριθμό. Τις περισσότερες τις ε, συμπεριέλαβα γιατί εξισορρόπησαν το κείμενο το βελτίωσαν. Συμφωνώ με τις περισσότερες τροπολογίες που προτείνονται στην παράγραφο α. Είναι οι 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12. Το περιεχόμενο των τροπολογιών δίνει μια πληρέστερη εικόνα της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσθέτει και άλλα στοιχεία που είναι στατιστικά χρήσιμα. Θεωρώ ότι οι τροπολογίες αυτές μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα συμβαστικό κείμενο. Δεν έχω καμία αντίρρηση τροπολογία 14. Επίσης, συμφωνώ με την τροπολογία 15 και την 17 που αφορούν στοιχεία που πραγματικά συμφωνώ ότι πρέπει να μας ανησυχούν. Οι τροπολογίες στην παράγραφο 2 κυρίως ασχολούνται με την ε, ολοκλήρωση της εικόνας της κατάστασης στα κράτη της ε, Ευρωζώνης. Τροπολογίες 18, 20, 21, 22, 23 και 24. Σημείωσα το αίσθημα ότι οι θετικοί δείκτες μπορεί να ε, εκφράζουν μια αύξηση της επισφαλούς εργασίας που πρέπει να καταπολεμηθεί. Όμως ε, θα ήταν ακριβές να πούμε ότι όλες οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι επισφαλείς. Πιστεύω ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα περισσότερα στοιχεία που αναφέρουν τροπολογίες που μόλις προανέφεραν σε έναν λογικό συμβασμό υποστηρίζω τις τροπολογίες που περιγράφουν τις τρομερά διαφορετικές καταστάσεις στα διάφορα κράτη-μέλη για τις τροπολογίες στην παράγραφο 3. Βλέπω να υπάρχει σημαντικός σκεπτικισμός όσον αφορά τα ενδεχόμενα αποτελέσματα των συστάσεων ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μπορώ να δεχθώ μια σειρά από τις αλλαγές που προτείνουν οι συνάδελφοι Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα και εδώ να επιτύχουμε συμβιβασμό. Συμφωνώ ότι πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στι ε, θέσει εργασία υψηλού επίπεδου, όπω αναφέρει η τροπολογία 54 για την παραγραφό 4. Καλωσορίζω τι τροπολογίε που καλούν να αυξηθεί η δημοκρατική λογοδοσία και η διαφάνεια, όπως η τροπολογία 59 Πολλές ε, πολύτιμες ιδέες προτάθηκαν για αυτή την παράγραφο, αλλά θεωρώ ότι ορισμένες πάνε κάπως υπερβολικά μακριά. Για παράδειγμα, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ε, κοινωνικών επιδομάτων δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Για την τροπολογία 64. Συμφωνώ ότι ένας κοινωνικός πυλώνας θα ήταν χρήσιμος, αλλά διαφωνώ ότι αυτός ο πυλώνας θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός της ε, ΟΝΕ θα έπρεπε να είναι παράλληλος προς την ΟΝΕ για τις τροπολογίες επί της παραγραφού 5 κυρίως θέλουν να, να, να απαλληφθεί η αναφορά στην ευελιξία μπορώ να το δεχθώ και μπορώ επίσης να δεχθώ να συμπεριληφθούν αναφορές στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στις θέσεις εργασίας ε, υψηλού επίπεδου. Για τι τροπολογίε 87 και 88 καταλαβαίνω τη σημασία της ε, σταθερότητας των τιμών, αλλά θα ήμουν επιφυλακτικό για το αν πρέπει να συμπεριληφθούν τέτοια μέτρα στις συνθήκε. Λοιπόν, προσβλέπω στι παρατηρήσεις των συναδέλφων μου και είμαι πεπισμένο ότι θα επιτύχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε συνένεση για να έχουμε μια ακριβή και ισορροπημένη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του, των σοσιαλιστών, Χαβιέ Λόπεθ. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κάσα για την εργασία του αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Είναι η πρώτη φορά που η Επίτροπή μας ε, κάνει τέτοια γνωμοδότηση και θα έπρεπε να το συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Θεωρούμε ότι ο συμβασμός είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για να εργαστούμε τις επόμενες εβδομάδες. Ε, η ομάδα μου δεν έβλεπε καθόλου να αντανακλώνται οι απόψεις της στο πρώτο κείμενο και πιστεύω ότι με τους συμβασμούς που προτείνονται σήμερα μπορούμε να έχουμε ένα πιο ισορροπημένο κείμενο για να εγκριθεί από την Επιτροπή μας και να είναι μια ισχυρή γνώμη που να βοηθήσει την εργασία του Κοινοβουλίου. Να σημειώσω τώρα ποιες ήταν οι κατευθυντήριες ε, γραμμές μας για την οικονομική και νομισματική πολιτική που ασκεί η ΕΚΟΥΤΟΥ από το 2013 και εντεύθεν. Πρώτον, η κατάσταση αγοράς εργασίας είναι πολύ ανησυχητική. Το μακροοικονομικό πλαίσιο είναι αρνητικό και θα συνεχίσει να είναι αρνητικό με βάση και τα στοιχεία του παρελθόντος θέρους. Αλλά ξέρετε από το 2013 αυξήθηκε η ανεργία και το 2014 διατηρήθηκε σε πολύ ψηλό επίπεδο και είναι πολύ άνηση ανεργία μεταξύ χωρών και ηλικιών. Βεβαίω. Έχουμε λιγότερη πίστη και λιγότερες επενδύσεις. Βεβαίως είναι πολύ χαμηλά τα επιτόκια, τα μείωσε το 2013, αλλά επαρκές δεν είναι αυτό, είναι προφανές. Χρειαζόμαστε πολιτικές πιο ε, ανορθόδοξες, λιγότερο συμβατικές. Να χρησιμοποιήσουμε, όπως θα ο και το ελικόπτερο. Υπάρχει ένα διαρθρωτικό πρόβλημα της ε, ΟΝΕ, πρέπει να ρυθμιστεί αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να δράσουμε μόνο επί της προσφοράς. Πρέπει βεβαίω να είναι λιγότερο επιθετική η δημοσιονομική πολιτική και η φορολογική πολιτική να έχουν δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτό το περιθώριο. Και για τη ζήτηση να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Αλλά όχι που να αυξήσουν την επισφάλεια, την ανισότητα. Γιατί υπάρχει κίνδυνο να αυξηθεί η επισφάλεια. Και αυτή η προσωρινή εργασία σημαίνει και περισσότερη ανασφάλεια. Εμένουμε δεν αναφέρεται στο συμβασμό Πρέπει να έχει λοιπόν διτή εντολή, να ελέγχει τις τιμές και να προωθεί την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και περισσότερη δημοκρατική λογοδοσία. Και κατά λίγο. η κίνδυνη για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι προφανής. Έχουμε το ενδεχόμενο αποπληθωρισμού και στασιμότητας. Κυκλική στασιμότητα που όλοι την ε, κατακρίνουν. Ποια είναι η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι να δώσουμε νομισματικά κίνητρα και φορολογικά κίνητρα για να αυξήσουμε, να τονώσουμε τη ζήτηση. Και δεύτερον, μεταρρυθμίσεις για να ευνοήσουμε περαιτέρω ανάπτυξη. Τα λέμε ήδη από καλοκαίρι, έπρεπε να το πει ο Τζάκσον Χολ για να το καταλάβουμε. Το αναφέρουν ε, τα βιβλία, τα πανεπιστημιακά για τη μακροοικονομία. Έχουμε τρία προβλήματα λοιπόν στην Ευρώπη. Πρώτον, δεν επαρκούν τα πολύ αδύνατα ε, νομισματικά κίνητρα, τα φορολογικά κίνητρα δεν έχουν προκύψει και τρίτον, χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις που επαρκώς, επαρκείς και αυτές δεν είναι. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Τριμπέσιος από το ECR έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και την ομάδα του για την πολύ καλή συνεργασία και την ιδιαίτερη προθυμία για την εξέβρεση συμβιβασμών. Και θεωρώ ότι στο μέλλον θα πρέπει να συνεργαστούμε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ομάδα του ECR, των συντηρητικών και των μεταρρυθμιστών. Θα καταλήξουμε σε ένα έγγραφο και θα βρούμε συνένεση. Εκ παραλλήλου θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία της πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα οποία η ομάδα μου και το κόμμα μου τα επικρίνει ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την ε, αναβολή χρεών στον ισολογισμό της ΕΚΤ. Δεν θα ευνοήσει αυτό τους φορολογούμενους και φυσικά ούτε πρόκειται να μειώσει τον αριθμό των ανέργων στην Ευρωζώνη. Σύμφωνο να συνεχίσει να παροτρύνει και να καλεί τα κρατημέλη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την διενέργεια των απαραίτητων διαθετικών αλλαγών στην αγορά εργασίας και είμαι αισιόδοξη για το μέλλον του εγγράφου αυτού και για την εξέβριση συμβαστικών λύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Χάρκιν από την Άλντε. Η κυρία Χάρκιν, παρακαλώ, από την ομάδα των φιλελευθέρων. Madam Harkin, she's... Oh, Then we'll go to the GUE group να περάσουμε στην ομάδα της ΓΚΟΕ. Ο κύριος Λέι Not uh, oh. Ούτε αυτός είναι εδώ. Α. Χαίρομαι, χαίρομαι, γιατί έτσι θα προλάβουμε. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στην διάθεσή μας. Στους πράσινους λοιπόν τώρα ο λόγος. Καρή Μαντελή. Όχι, ούτε αυτή. Ε, τότε, από το EFTD, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κάζα για την εργασία, για τη δουλειά του. Υπάρχει ένα λίγο πιο ανοιχτό πνεύμα σε ό,τι αφορά τις επιθυμίες που εκφράσαμε Στην αρχή το κείμενο δεν μας ε, φαίνονταν καθόλου ισορροπημένο. Δεν συμφωνούσαμε ιδιαίτερα. Τώρα βλέπουμε ότι στην πορεία των διαπραγματεύσεων, μέσω των τροπολογιών, λαμβάνονται υπόψη και τα δικά μας τα στοιχεία που μας απασχολούν ιδιαίτερως. Υπάρχουν ε, τροπολογίες τις οποίες και καταθέσαμε οι οποίες είναι βασικές για μας, θεμελιώδους σημασία, γιατί με αυτές τις τροπολογίες υπογραμμίζεται η οικονομική κατάσταση, η κατάσταση στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά αυτά που ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Ένα σημαντικό σημείο το οποίο και θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι το σύμφωνο σταθερότητας το 3% και ο σχετικός περιορισμός. Αυτό πραγματικά για μας είναι κάτι το απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Αν ένα κράτος δεν έχει δυνατότητα να επενδύει δεν έχει δυνατότητα να βοηθήσει την πραγματική οικονομία. Οι νομισματικές ροές δεν μπορούν να κινούνται μόνο προς τις τράπεζες. Πρέπει να κινούνται και από τις τράπεζες προς την πραγματική οικονομία. Ιδιαίτερος προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους ιδιώτες. Ιδάλλως δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ύστερα, Άλλο ένα σημαντικό σημείο για μας είναι η τροπολογία υπαριθμών 12. όπου το θέμα είναι η ανεργία. Δεν παρουσιάζεται με ισόρροπο τρόπο όμως η κατάσταση. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να θίξω το εξής ε, θέμα. 7,7 άπτια στη Γερμανία 57,3% η ανεργία στην Ελλάδα. Είναι σαφή τα αριθμητικά στοιχεία και μιλάνε από μόνα τους νομίζω. Ε, Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα θέματα αυτά, να μιλάμε για την ε, το δημοκρατικό ρόλο, τον διαφανή δημοκρατικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ευθύνη που φέρει. Θα πρέπει λοιπόν να πετύχουμε τη διαφάνεια αυτή. Πάρα πολλά σημεία υπάρχουν που είναι κρίσιμα. Η γνωμοδότηση δεν είναι ισόρροπη. Είναι πολύ λίγα τα αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται. Θέλουμε να υπάρχει αναφορά στην αύξηση της απασχόλησης στις χώρες που δεν έχουν το ευρώ. Γιατί δεν λέμε ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν στα χώρα, στις χώρες που έχουν εισαγάγει το ευρώ. Κοιτάμε και βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση στις ε, χώρες αυτές. Πολλά σημεία λοιπόν μας απασχολούν ιδιαίτερα, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχει μια διάθεση συμβιβασμού. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο, ο κύριο Κάζα για να συνοψίσει. Εν συντομία να απαντήσω στου συναδέλφους σε ό,τι αφορά την ανάλυση των τροπολογιών. Να σα ευχαριστήσω. Να σα ευχαριστήσω και για το πνεύμα συνεργασία, το οποίο και ελπίζω να παραμείνει, να συνεχιστεί τι επόμενε ημέρε, προκειμένου να βρούμε κοινό έδαφο και να παράγουμε τελικά μια ακριβή και ισορροπημένη γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Κάζα και όλους τους υπόλοιπους. Πρώτη και δεύτερη Δεκεμβρίου στην Επιτροπή ε, Απασχόλησης. Στις 8 ε, Δεκεμβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή Οίκων και το Φεβρουάριο του επόμενου έτους θα πάει στην Ολομέλη το θέμα. Και τώρα να περάσουμε στο 8 της ημερησίας διάταξης. Ζητήσαμε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Απασχόλησης τη διενέργεια μιας μελέτης για τα άτομα με αναπηρία σε ό,τι αφορά την εύλογη προσαρμογή και τον καθολικό σχεδιασμό, σε ό,τι αφορά τις σχετικές επενδύσεις. Επτά άτομα συμμετείχαν στην κατάρτιση της έρευνας αυτής. Έχουμε τον κύριο Κουέντιν Λιζέ μαζί μας και τον κύριο, και Χάρπερ που εκπροσωπούν και τους επτά συγγραφείς της μελέτης αυτής και θα μας παρουσιάσουν εν συντομία τα πορίσματα της έρευνας ε, τα οποία και τους ζητήσαμε να ερευνήσουν. Ο κύριος Λίζε έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ με τον κύριο Χάρπερ Είμαστε από την εταιρεία Optimum Matrix και μας ζητήθηκε να διενεργήσουμε αυτή τη μελέτη, όπως είπε η Πρόεδρος, και να παρουσιάσουμε τα πορίσματα. Μιλάμε λοιπόν για λογισμένες προσαρμογές σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρίες, σε ό,τι αφορά το κόστος και την απόδοση των επενδύσεων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να χαρτογραφήσουμε την κατάσταση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να βρούμε κάποια ενδιαφέροντα παραδείγματα σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που απαντώνται, σε ό,τι αφορά τα διδάγματα που μπορούμε να εξαγάγουμε, σε ό,τι αφορά το κόστος και την απόδοση των επενδύσεων για κάποιες από τις αποφάσεις των νομοθετών. Μάλιστα. Η παρουσίασή μου θα είναι αυτή λοιπόν δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο φαίνεται. Να σας παρουσιάσω εν συντομία λοιπόν την παρουσίαση. Μιλάμε το κόστος και, για το κόστος και την απόδοση των επενδύσεων για τα άτομα με αναπηρία σε ό,τι αφορά τα προστατευόμενα εργαστήρια και τις λογισμένες προσαρμογές. Οι λογισμένες προσαρμογές λοιπόν κοιτάμε και το καθολικό σχεδιασμό. Θεωρούμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει και ανάγκη ομαδοποίηση των δύο κλάδων αυτών. Και κοιτάξαμε και τις γενικότερες πολιτικές, γιατί οι ορισμοί στα διάφορα κράτη-μέλη είναι διαφορετικοί. Και είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε τι θεωρείται λελογισμένη προσαρμογή. Θα σας το εξηγήσω λοιπόν πιο λεπτομερώς. Εστιαστήκαμε σε έξι κράτη-μέλη. Βέλγιο, Γερμανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία και Ισπανία. Και κάναμε λοιπόν ε, διαφορετικές οικονομικές αναλύσεις. Κάποιες ήταν αναλύσεις ε, ε, και δαπάνης. Κοιτάξαμε το, κοιτάξαμε το γερμανικό σύστημα ποσοστώσεων και την αλλαγή του συστήματος ποσοστώσεων και τα πορίσματα το 2000. Το, σχέδιο, το νομοσχέδιο για την ε, διακριτική μεταχείριση των ε, αναπηριών στον Εμένο Βασίλειο, στην Ουγγαρία, το ένα πρόγραμμα ESF ε, στη Λιθουανία, Towards Work ονομάζεται, και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια διαφορετική προοπτική κοιτώντα ε, την υποστηριζόμενη απασχόληση στις ΕΠΑ και κάναμε αναθεώρηση διάφορων μελετών που ονομάζονται Individual Placement Surveys. Για να σας δώσω την οικονομική διάσταση, να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο Γκάρετ. Ευχαριστώ. Όπως είπε ο Κουέντιν, η μεθοδολογία που χρησιμοποίησαμε είναι μια ανάλυση κόστους και ωφέλους. Να σας εξηγήσω λοιπόν τι προσπαθούμε να πετύχουμε στην προκειμένη περίπτωση. Όπως λέει και ο ίδιος ο τίτλος, Σκοπός είναι να κοιτάξουμε διάφορες παρεμβάσεις, να καταλάβουμε ποιο κόστος συνεπάγονται σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους και να τα συγκρίνουμε με την αποτελεσματικότητα και πώς ε, επηρεάζουν τους στόχους που θέσαμε στην αρχή. Ο ρόλος λοιπόν της ανάλυσης αυτής είναι να συγκρίνουμε το κόστος και το όφελος με ένα κοινό μορφότυπο σε χρηματικούς όρους και να δούμε κατά πόσον οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ε, αξίζουν τον κόπο και είχαν απόδοση της επένδυσης. Και συχνά στις περιπτώσεις αυτές, σε κάποιες περιπτώσεις ο αντικτύπος δεν, είναι, δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κοιτάξουμε κατά πόσο ήταν σημαντικό ο αντίκτυπο σε περίπτωση που δεν μπορούσαμε να θέσουμε ένα πόσο. Ένα άλλο θέμα σε αυτέ τι αναλύσει είναι το θέμα τη προπτική. Θα δείτε στην έκθεση ότι ο αριθμό ε, των προοπτικών που περιλαμβάνεται είναι διαφορετικός. Κοιτάμε από οπτική του ατόμου, κοιτάμε από την οπτική γωνία των ε, δημόσιων αρχών, κατά πόσον υπάρχει βελτίωση σε ό,τι αφορά την απασχόληση ή μπορούμε να κοιτάξουμε και την οπτική γωνία την κοινωνική. Στο σύνολο της κοινωνίας, κατά πόσον υπάρχει ε, γενικότερη ποιότητα ζωής, ικανοποίηση. Είναι δύσκολο. Κάναμε λοιπόν μία απόπειρα να ποσοτοκοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία. Και τέλος, κοιτάμε το πόσο καλά μπορούμε να βρούμε το αίτιο και το αιτιατό για να δούμε κατά πόσον αυτό που κάναμε επηρέασε και έφτασε και ε, βοήθησε στην επίτευξη του στόχου που προσπαθούμε να πετύχουμε. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα θέματα μεθοδολογικών αλλαγών Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γκάρατ. Το λόγο έχει πάλι ο κύριος Λιζέ. Κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, η πρώτη πρόκληση δεν ήταν η πρόκληση, αλλά το θέμα το οποίο εξετάσαμε, το ποσοστό απασχόλησης των αναπήρων διπλό σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ως οικονομολόγοι λοιπόν κοιτάμε καταρχάς τον ορισμό των ε, αναπήρων στις διάφορες χώρες. Υπάρχει ο κοινωνικός, ο ιατρικός όρος, ο ιατρικός ορισμός λέει ότι ένα άτομα δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, Είναι ο κοινωνικός ορισμός ε, εστιάζεται πιο πολύ στην κοινωνία, στο περιβάλλον και λέει ότι ο κόσμος είναι σε θέση αναπηρίας ε, λόγω του τρόπου με τον οποίο ζούμε και όχι τόσο πολύ λόγω των σωματικών του αναπηριών. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν αυτή η διάκριση. Κοιτώντας το όλο θέμα αυτό των ε, αναπηριών, γιατί υπάρχουν και πολλές διαφορετικές αναπηρίες, ε, ψυχικής υγείας, ε, σωματικής υγείας. βάση λοιπόν των διαφορών αυτών, καταλήξαμε γρήγορα στο συμπέρασμα ότι σε όλα τα κρατημέλη οι ίδιοι όροι δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα και ο ορισμός, οι ορισμοί δεν είναι ξεκάθαροι. Είναι δύσκολο λοιπόν να βρούμε και να καταλήξουμε το τι εννοείται σε κάθε κράτος μέλος. Προσπαθήσαμε όμως να το κάνουμε αυτό. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τα προστατευόμενα εργασίρια δεν υπάρχει κοινό ορισμό των προστατευόμενων εργαστηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούσαμε ότι υπήρχε ένα κοινό ορισμό μέρη που απασχολούν άτομα με αναπηρίε. Άτομα με αναπηρίες συνεργάζονται σε προστατευόμενο περιβάλλον από άλλου είδους εργαζομένων όταν προσπαθήσαμε να τα θέσουμε όλα αυτά σε ένα διάγραμμα, διαπιστώσαμε ότι αυτά τα εργαστήρια έχουν συχνά διάφορους σκοπούς. Σε κάποια κράτη-μέλη σκοπός είναι να βοηθήσει τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Και είναι μία εναλλακτική στην, ε, αν θέλετε, στην ε, περίθαλψη η μετάβαση προς την απασχόληση φαίνεται να είναι πολύ πιο σημαντική, αλλά προκάλεσε και, προκαλεί και κάποια προβλήματα. Αυτό που προσπαθούμε να καταδείξουμε είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά διαφορετικοί ορισμοί των παραδοσιακών και των μεταβατικών εργαστηρίων, θεωρούμε ότι όλα υπάγονται στον ίδιο άξονα σε ό,τι αφορά την ανάλυση κόστους και ωφέλους. Κοιτάξαμε την καθαρά οικονομική διάσταση και είδαμε ότι στην περίπτωση του Σίβιταντ, ενός ουγγρικού εργαστηρίου, δεν υπήρχε απόδοση της επένδυσης απαραίτητα, γιατί τα χρήματα που θα πάνε σε κυβέρνηση ήταν 20 λεπτά ανά ευρώ που δαπανόταν. Το πραγματικό ερώτημα είναι αυτό πρέπει να κοιτάμε, γιατί η απόδοση των επενδύσεων, όπως είπε ο Γκάρετ, δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί απαραίτητα. Η εναλλακτική λύση θα ήταν να μην εργάζονται οι άνθρωποι αυτοί, αλλά να είναι σε ένα νοσοκομείο, σε κάποιο καθεστώς φύλαξης, να απασχολούν τις οικογένειές τους. Ένα άλλο θέμα το οποίο και διαπιστώσαμε είναι ότι στα μεταβατικά εργαστήρια που προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο να κινηθεί προς την ελεύθερη αγορά εργασίας φαίνεται ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ατόμων που περνούν από τη μεταβατική αυτή φάση εργαστηρίων στην αγορά εργασίας. 3% νομίζω. Νομίζω ότι αυτό το ποσοστό χρησιμοποίησε και η Επιτροπή σας ε, πέρσι. Το ποσοστό αυτό βαθίστηκε σε μία μελέτη του 2009. Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι, ακόμα κι αν φτάσουν στο καθεστώς της ε, απασχόλησης, η εργασία αυτή μπορεί να είναι πολύ προσωρινής διάρκειας. Ε, ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα έχουμε από τη Σουηδία. Για εργαζόμενους σε τέτοια εργαστήρια που περνούν ε, στην κανονική αγορά εργασία, αλλά έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο εργαστήριο. Σάμχαλ ονομάζεται το παράδειγμα από τη Σουηδία. Να δούμε λοιπόν τώρα τους όρους και πώς ορίζονται. Τι είναι οι λελογισμένοι, εγκαταστάσει. Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις στην αγορά στη θέση, στην ε, εκάστοτε εργασία. Να μην υπάρχει δυσανάλογο βάρος που να επιβαρύνει τον εργοδότη. Οι λελογισμένες λοιπόν εγκαταστάσεις ε, μπορεί να είναι από τη ράμπα για το καροτσάκι, αλλά μπορεί να είναι και κοινωνική υποστήριξη για τα άτομα με ζητήματα για την ε, ψυχική τους υγεία, για να μπορούν να διατηρήσουν τη θέση εργασίας. Και όπως ανέφερα προηγουμένως, αυτό συνδέεται με τον καθολικό σχεδιασμό και ελπίζω να το βλέπετε αυτό από την εικόνα σε ό,τι αφορά και τον κοινωνικό ορισμό των αναπηριών. Αν ξεκινήσουμε να οικοδημούμε ένα περιβάλλον γενικότερα που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες, θα μειώσουμε την ανάγκη να γίνονται εκ των υστέρων αλλαγές στην, ε, στο χώρο εργασίας. Μία ράμπα λοιπόν ε, που μπορεί να προσθεθεί ή δεξιά στην εικόνα βλέπετε πως μπορεί να ενσωματωθεί η ράμπα από την αρχή. Νομίζω ότι για πρώτη φορά ε, χρησιμοποιήθηκε η έννοια αυτή στις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Και βλέπουμε λοιπόν αυτό το, αυτή την αρχή του καθολικού σχεδιασμού σε διάφορες ε, τεχνολογίες. Κοιτώντας τώρα λοιπόν την απόδοση των επενδύσεων. Βλέπουμε ότι πολλά, πολύ λίγα έχουν γίνει για ε, λογικές εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρίες. Ένα από τα ποσοστά που συχνά αναφέρονται είναι το ποσοστό 1 προς 48. 1 ευρώ για κάθε 48 ευρώ που επενδύονται. Αλλά αυτό το στοιχείο, αυτό το ποσοστό, αυτή η αναλογία στον Ομένο Βασίλειο είναι πολύ αμφίβολη. Τώρα μάλλον ισχύει το 1 προς 18, 1 ευρώ προς 18. Έχουν γίνει κάποιες δαπάνες, ε, ε, κάποιες μελέτες στην ε, Ολλανδία που φαίνεται ότι καταδεικνύουν ότι υπάρχει απόδοση της επένδυσης. Και τέλος κοιτάμε τις εναλλακτικέ υπηρεσίες για την αγορά εργασίας. Είναι ένας τομέας που διαιρείται σε αυτούς τους τέσσερις κλάδους που βλέπετε. Καταρχάς, ε, ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, κάποιες θετικές δράσεις, εκπαίδευση, καθοδήγηση, συμβουλευτική για να βοηθηθούν τα άτομα αυτά να βρουν ε, δουλειά. Για τα προγράμματα εργασίας στη Λιθουανία, όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι ενδιαφέρον το έργο αυτό και ουσιαστικά ε, σας είπα ότι χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το ESF. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βοηθά τους κοφούς να βρουν θέση εργασίας, εκπαιδεύοντας άτομα που θα τα βοηθήσουν να βρουν απασχόληση, που θα κατανοήσουν τις ανάγκες τους και που θα μπορέσουν να το μεταβιβάσουν αυτό ως μήνυμα στον ενδεχόμενο εργοδότη. Ένα από τα θέματα που ανέκυψε είναι ότι παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε από το από το 2009 μέχρι το 2012, τα άτομα που εκπαιδεύτηκαν συνεχίζουν να εργάζονται και άρα ο είναι πολύ μεγαλύτερο. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, υπήρχε απόδοση τη επένδυσης, αλλά πολύ περισσότερη μεγαλύτερη απόδοση ήταν σε μακρυπρόθεσμο επίπεδο. Δεύτερον, ε, παθητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας. Αυτό είναι λίγο πιο αμφιλεγόμενο. Περιλαμβάνει μέτρα, για παράδειγμα, για την αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος, ε, επιδοτήσεις ε, μισθού, ε, βοήθεια προς τους, εργαζο... προς τους εργοδότες για να απασχολούν ή να κρατούν σε απασχόληση ανάπηρα άτομα. Το βασικό θέμα εδώ φαίνεται ότι είναι ότι τα άτομα με αναπηρία θεωρούν ότι είναι στιγματισμένα αν απασχολούνται μέσω τέτοιων πολιτικών αγοράς εργασίας. Γιατί οι μελέτες καταδεικνύουν ότι τα άτομα με αναπηρία που απασχολούνταν υπό τέτοιο καθεστώς έχουν την αίσθηση ότι για αυτόν τον λόγο τους απασχολούν και όχι για τα πραγματικά τους προσόντα και για την ικανότητά τους να κάνουν τη δουλειά τους. Τα γενικότερα μέτρα τα οποία εξετάσαμε και εδώ θα επισέλθω σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας γιατί κάναμε και ανάλυση κόστους ωφέλους έχουν θετικό αντίκτυπο. Είναι όμως ευρείες πολιτικές, πολύ ευρείες, που δεν αφορούν ειδικότερα την απασχόληση, αλλά γενικότερα. Κοιτάξαμε λοιπόν τις διακρίσεις για λόγους ε, αναπηρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο Γκάρεθ μπορεί να σας πει περισσότερα για την οικονομική ανάλυση για το θέμα αυτό. Αλλά από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που εγκρίθηκε το συγκεκριμένο νομοθέτημα παρά αυτό που θα θεωρούσαν προφανές θεωρείται ότι 180.000 άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν βρει δουλειά και αυτό δεν ωφελεί μόνο αυτούς τους εργαζόμενους σημαίνει ότι το 2013 υπήρξε μία αύξηση 361 εκατομμυρίων ε, λιρών ακαθάριστου εισοδήματος, κάτι το οποίο είχε βεβαίως και ε, επιπτώσεις σε αυξημένα φορολογικά έσοδα και έσοδα για την κοινωνική ασφάλιση. Μετά εξετάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα, δηλαδή ποσοστώσεις. Είχαμε τέτοιες ποσοστώσεις σε 21 κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα εξετάσαμε την περίπτωση της Γερμανίας, γιατί είχαμε στοιχεία πιο προσβάσιμα. Διαπιστώσαμε ότι το 2000 άλλαξε το γερμανικό σύστημα ποσοστώσεων. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Μειώθηκε μεν η ποσόστοση, αλλά η δομή των ποινών και κυρώσεων τροποποιήθηκε και περιμέναμε ότι θα είχε αρνητικό αποτέλεσμα η μείωση των ποσοστώσεων, αλλά η αλλαγή στην δομή κυρώσεων τελικά είχε πολύ εντονότερο αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή της δομής. Σημαίνει πως είναι πολύ πιο ακριβό για τους εργοδότες να μην πληρούν την ποσόστοσή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ότι το ενδεχόμενο απασχόλησης ε, ατόμων με ειδικές ανάγκες αυξήθηκε ε, μεταξύ 2,2 και 3,5% ενώ ήταν πολύ μικρή η αλλαγή όσον αφορά το κόστος των κυρώσεων. Συνολικά, τι διαπιστώσαμε. Τι θα προτείναμε. εγώ είμαι περισσότερο αποτιμητής. Ο Γκάρεθ είναι οικονομολόγος. Στην ομάδα μας έχουμε αποτιμητές, οικονομολόγους και ε, εκφραστές πολιτικής. Ένα πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν σαφείς και συγκρίσιμοι ορισμοί. Αυτό δυσχεραίνει πολύ την συγκριτική έρευνα μεταξύ των κρατών μελών. Σε σχέση με αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Αλλά ιδιαίτερα χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες και αναλυτικές επιστημονικές μελέτες, πανεπιστημιακές μελέτες για το πόσο κοστίζει και πόσο αποδίδει τελικά αυτή η πολιτική. Έχουμε μια συγκεκριμένη ε, μελέτη για άτομα με προβλήματα ε, διανοητικής υγείας που ξεκίνησε στι Ηνωμένε Πολιτείε και έχει εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα στην Ένωση είχαμε αυτή τη ε, μελέτη σε έξι διαφορετικές πόλεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά και σε κάθε ε, τέτοια μελέτη είχαμε μία ομάδα ελέγχου και μία ομάδα ατόμων που είχαν τα προβλήματα και αυτό απέδειξε ότι χρειάζεται τέτοια μελέτη και τέτοιες έρευνες Επίσης είναι πολύ θετικέ επιπτώσεις στην κοινωνική αντίληψη για τα άτομα αυτά. Και αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η διάθεση να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά. Αυτό είναι πολύ πιο θετικό από απλώς επιμέρους αλλαγές. Και επίσης, κάτι που δεν ήταν εντελώ μέσα στη μελέτη, διαπιστώσαμε ότι πολύ συχνά αν υπάρχει εύλογη προσαρμογή χρηματοδοτούμενη από τις κυβερνήσεις μέσω των εισόδων των εσόδων συγγνώμη, από τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις εταιρείε που δεν πληρούν τις ποσοστώσεις αυτή η αντίληψη δηλαδή όχι μόνο αυτά, αυτά τα χρήματα αλλά τα χρήματα από τα πρόστιμα για παράβαση της εργασιακής νομοθεσίας είναι χρήσιμα, βοηθάνε, βοηθάνε για να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα προστατευόμενα εργαστήρια και τις εύλογες προσαρμογές. Και επιπλέον το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να τονίσουμε ότι έχει βοηθήσει πολύ σε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την προσοχή σας και ε, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις φυσικά. Θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι? Όχι. Ο κύριος Χάουιτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταπληκτική μελέτη και είναι πολύ καλό που βλέπουμε και τις λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσαμε να βρούμε οικονομικά επιχειρήματα ώστε να έχουν ισότιμη μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας η ΑΜΕΑ. Μιλήσατε για τις εύλογες προσαρμογές ε, και νομίζουν όλοι ότι μιλάμε για τα σπίτια. Δυσκολεύονται και οι διερμηνείς, εξάλλου. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για προσαρμογές, ειδικέ υπηρεσίες στήριξης στο χώρο εργασίας. Η όρος accommodation λοιπόν στα αγγλικά έτσι πρέπει να ερμηνευτεί. Ποιες προσαρμογές γίνονται στο χώρο εργασίας. Άρχισα με τα ορολογικά αλλά ε, λύσαμε το μισό πρόβλημα. Νομίζω αν όλοι ξέρουν περί τίνο πρόκειται όταν συζητάμε. Ε, ποιες ερωτήσεις ήθελα να κάνω εγώ. Πρώτον, το παλαιό μοντέλο, μιλήσατε για το κοινωνικό μοντέλο για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες και υπήρχαν κάποια εργαστήρια, κάποια καλά, ε, κάποια πάλι όχι. Και ε, σημειώθηκε μια αλλαγή. Βελτιώθηκαν οι συνθήκες ε, στα προστατευμένα εργαστήρια, ούτως ώστε να δίνουν τις καλύτερες, τις βέλτιστες εργοδοτικέ πρακτικέ, αλλά πέραν από αυτού Πέραν από αυτό, υπήρξε καλύτερη υποστήριξη προς ε, τους ΑΜΕΑ μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Αυτή η τάση προς μεγαλύτερη υποστήριξη διαπιστώθηκε στις χώρες που μελετήσατε. Δεύτερον, σύμβαση του ΟΗΕ για τους ΑΜΕΑ. στην Ευρώπη και στον κόσμο υπάρχει μια δυναμική ε, υπέρ των και αναρωτιέμαι αυτοί που εκπονούν την πολιτική χρησιμοποιούν τη σύμβαση του ΟΗΕ κυρίως στα πλαίσια της απασχόλησης των ΑΜΕΑ ή όχι. Τρίτον, η οικονομική επίπτωση της των πολιτικών λιτότητας. Είναι ξεκάθαρο, έτσι δεν είναι, ότι έπεσαν θύματα η ΑΜΕΑ και έχουν μεγαλύτερες ε, πιθανότητες να παραμείνουν εκτός αγοράς εργασίας ή να μην έχουν τις υπηρεσίες που δικαιούνται. Δεν μπορεί να ασχολούμαστε με αυτή τη μελέτη και να μην αναρωτηθούμε κατά τη διάρκεια της δουλειάς σας τι σχετικό διαπιστώσατε. Εγώ κάνω και μια σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο και μια μελέτη που έγινε με αναπηρία έχετε διπλάσιες ε, πιθανότητες να είστε άνεργος. Υπάρχει έκθεση του ΩΣΑ, το ίδιο ισχύει για την αποζημίωση. Τα στοιχεία είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο και δείχνει ότι ε, ε, περικόπτηκε ε, τελείω ε, ο προπολογισμό, ο δημόσιο προπολογισμό για την υποστήριξη των ΑΜΕ από το 1,48 πέρασαμε στο 1,8. Είναι εντελώ αντιπαραγωγικέ οι περικόπε των δαπανών. Το 35% των δικαιούχων αυτού του προγράμματος ήταν αμαία, είχαν χρόνιες παθήσεις και τώρα, όταν ήταν το κόμμα μου στην κυβέρνηση και τώρα πλέον έχουμε περάσει στο 15% ε, και σίγουρα σοκάρουν αυτά τα στοιχεία. Ε, εγώ θέλω να ξέρω, πέρα από τον νόμο Βασίλειο, τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τι είδατε εσείς ε, στη μελέτη σας. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο και στην κυρία Πλουρατού και θα απαντήσουμε μαζί στις ερωτήσεις. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κι εγώ για τη μελέτη. Ευχαριστώ την Διεύθυνση Μελετών για την σφαιρική της προσέγγιση. Η προσέγγιση σας είναι ολιστική και πραγματεύεστε γενικότερα το ζήτημα της ε, στήριξης ε, των ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας. Ε, νιώθω ευγνωμοσύνη προς αυτούς που ζήτησαν την εκπόνηση αυτής της μελέτης στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Η σημερινή συνεδρίαση είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε για να συζητήσουμε το, τη μελέτη σας. Είναι αρκετά διεξοδική η μελέτη και περίπλοκο το θέμα της. Ε, η μελέτη προς το παρόν είναι διαθέσιμη στα αγγλικά μόνο. Γι' αυτό και δεν μπόρεσα να τη διαβάσω και να την αναλύσω. Δεν είμαι η μόνη νομίζω. Γι' αυτό ε, ήθελα να πω σε σχέση με την αυριανή προθεσμία για την υποβολή σχολείων ότι δεν είναι ρεαλιστικό, δεν έχουμε χρόνο για να υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας. θα πρέπει να ισχύσουν τα ίδια πρότυπα όπως αυτά που ακολουθούμε για τις εκθέσεις. Η μεθοδολογία μας είναι τέτοια ώστε χρειαζόμαστε ένα μήνα περίπου για να συμβουλευτούμε τους εμπειρογνώμονες και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Και είμαι σίγουρη ότι αυτή η μελέτη θα είναι σημείο αναφοράς και πολλοί θα παραπέμπουν σε αυτή, όχι μόνο για τη δική μας δουλειά, αλλά και για πολλούς άλλους ερευνητές. Θα είναι πηγή έμπνευση η έκθεσή σας. Θα συζητηθεί επίσης στα Εθνικά Κοινοβούλια. Λοιπόν, δοθεί τη σημασία, της κύριας σημασίας αυτής της έκθεσης είναι απαραίτητο να πηχεί την πραγματικότητα στα στοιχεία της έκθεσης θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι χρήσιμο εργαλείο για τη δουλειά μας αυτή η έκθεση. Θα ήθελα να εκφράσω μια γενική φύση αμφιβολία σε αυτό το στάδιο της συζήτησης. Εγώ πιστεύω πως στην έκθεση δεν απηχούνται ικανοποιητικά τα επιτεύγματα και τα απορίσματα της κοινή έκθεσης Παγκοσμίου ε, Οργανισμού Υγείας εκπαιδεύω το 2011 Γίνεται μια σε αναφορά στην έκθεση, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται έτσι αυτή η αναφορά. Δεν αναφερόμαστε σε αυτούς που την εκπώνησαν, δεν δίνονται αρκετές πληροφορίες για το περιεχόμενο της έκθεσης. Φαντάζομαι ότι έχετε ακολουθήσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. και ότι βασιστήκατε σε κάποια κριτήρια. Επιλέξατε μία ομάδα κρατών μελών. Λυπούμε που η Πολωνία δεν συγκαταλέγεται στις χώρες που διαλέξατε. Ε, παρομοίως, δεν υπάρχουν σχόλια πολωνών εμπειρογνωμόνων στην έκθεσή σας. Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι είναι πολύτιμη η έκθεση που συντάξατε και συναποτελείται από τα βασικότερα σημεία που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, ούτω ώστε οποιοδήποτε πολιτικός να μπορέσει να λάβει αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα, την κατάσταση και να μπορέσει να διαμορφώσει γνώμη και να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις για την εκπόνηση πολιτικής. Απευθύνω λοιπόν έκκληση Παρακαλώ να μας δοθεί αρκετός χρόνος για να μελετήσουμε διεξοδικά την έκθεση, να υποβάλουμε τα σχόλιά μας. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Άνταμ Κόσα, μάλλον σε αυτό που πιστεύει ο κύριος Άνταμ Κόσα, ε, συμφωνεί μαζί μου ότι πρέπει να παραταθεί η προθεσμία για την υποβολή των σχολείων των βουλευτών. Κυρία Ολσκο, ευχαριστούμε. Μιλήσατε για την έλλειψη μεταφράσεων της έκθεσης και για την ε, προθεσμία. Το τμήμα μελετών θα ασχοληθεί με το θέμα. Έχει 232 σελίδες η έκθεση. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σίγουρα το τμήμα μελετών θα επανέλθει και θα μας κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς που επιθυμούν να εμβαθύνουν να μελετήσουν την έκθεση και να υποβαλούν δικές τους ε, παρατηρήσεις. Επανέλθει λοιπόν το τμήμα μελετών. Αυτή είναι η πρώτη σύντομη απάντηση στις ε, ερωτήσεις του κυρίου Πλούρα. Έχουμε έναν ροκά στη Σουηδία που ονομάζεται Πλούρα συνονόματος. Θα, ήθελε, θα θέλατε να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Θέλω να απαντήσω και σε κάποια άλλα ερωτήματα του κ. Χάιτ μεταξύ άλλων σε ποιο βαθμό μας ρώτησε υπήρξε αλλαγή στροφή στην πορεία που ακολουθούμε για τα προστατευμένα εργαστήρια. Όπως σωστά είπε, δύο είναι τα ζητήματα. Πρώτον, ο στόχος των εργαστηρίων και εκεί φυσικά τίθεται ζήτημα συνθήκων και προτύπων λειτουργίας των εργαστηρίων σε κάποια κράτη-μέλη θεωρούνται εργαζόμενοι αυτοί που απασχολούνται στα εργαστήρια αλλά όχι σε όλες χώρες. Υπάρχουν διάφορα στρώματα προβλημάτων που διαπιστώσαμε μέσα στην έκθεση. Αυτό είναι ένα στρώμα. Μπορούμε να συντάξουμε άλλες δέκα εκθέσεις ε, εξίσου ογκώδης ε, για να αναφερθούμε σε όλα αυτά που διαπιστώσαμε. Για τη σύμβαση του ΟΗΕ τώρα, για τους ΑΜΕΑ, Στη σελίδα 35 κάνουμε αναφορά και στη σύμβαση και ε, στο προαιρετικό πρωτόκολλο. κάποια κράτη το έχουν υπογράψει, αλλά δεν το έχουν επικυρώσει, άλλοι το έχουν επικυρώσει. Ε, είναι το γενικότερο θέμα αν μετά την ε, έγκριση νομοθεσίας έπεται εφαρμογή, σωστή εφαρμογή. Και αυτό με φέρνει και στο σημείο που θα σχολιάσει ο συνάδελφός μου για την οικονομική διάσταση του ζητήματος και την οικονομική κρίση. Τα μέτρα που εξετάσαμε χαρακτηρίζονται από τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κάλυψε ένα πολύ μεγάλο κενό χρηματοδότησης από πλευράς των κρατών μελών ε, δηλαδή χρηματοδότηση που δεν προσφέρουν τα κράτη-μέλη λόγω της οικονομικής κρίσης. Υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα αφήσω τον Κάρθ να μας μιλήσει γι' αυτό και μετά θα επανέλθω στις δικές σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ. ως προς ε, τις πολιτικές λιτότητες και τον οικονομικό αντίκτυπο. έχει μια συγκεκριμένη αναφορά στις επιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έγινε ανάλυση στα οικονομικά κεφάλαια για ε, το νομοσχέδιο για τα άτομα με αναπηρίες. Ε, για μια δεκαετία ασχοληθήκαμε με αυτό το ζήτημα. Έγινε ανάλυση της κατάστασης, όμως το γενικότερο ζήτημα ε, των μακροοικονομικών, των επιπτώσεων της μακροοικονομικής ε, πολιτικής ε, στην αγορά εργασίας είναι ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής ανάλυσης για την κατανομή των επιπτώσεων και βάσει της τεκμηρίωσης που έχουμε προκύπτει ότι μεγαλύτερος αντίκτυπος παρατηρείται στους τομείς όπου υπάρχει η πιο ισχυρή μετάβαση. Δηλαδή, εκεί όπου επιχειρήσεις, δραστηριότητα των επιχειρήσεων επηρεάζονται από την οικονομική συγκυρία. Δεν έχω τα στοιχεία μαζί μου, αλλά μπορώ να σας πω ότι υπάρχει δυσανάλογα μεγάλος αντίκτυπος στις επιχειρήσεις ή σε, εκείνες τις, σε εκείνους τομείς αγοράς εργασίας που επηρεάζονται ούτως ή άλλως περισσότερο από την οικονομική κρίση. Ευχαριστούμε. Δεν μπορώ να σχολιάσω ούτε την προθεσμία ούτε το θέμα των γλωσσικών μεταφράσεων, κύριε Πλούρα αλλά μας ρωτήσατε γιατί όχι την Πολωνία. Έξι ε, κράτη-μέλη επιλέξαμε, αναγκαστικά 22 μένουν απ' έξω. Όλοι φυσικά θα ήθελαν να είναι μέσα στην έκθεση. Προσδοποιήσουμε βέλτιστες ε, πρακτικές και ε, καλή σχέση κόστος-οφέλους. Ο στόχος δεν ήταν περιστατωμένα και πλήρως να καταγράψουμε την κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αλλά αναφερόμαστε στην Πολωνία σε διάφορε σημεία και αν μεταφραστεί η έκθεση στα πολωνικά θα το διαπιστώσετε. Ε, είπατε ότι δεν αναφερθήκαμε σε όλη την βιβλιογραφία ε, στην οποία παραπέμπουμε και μιλήσατε για την έκθεση του ΠΟΗ. Ε, ο στόχος ήταν να ασχοληθούμε με την οικονομική ανάλυση γιατί κάνουμε αναχώρα μελέτες θα σας απαντήσω ότι αν είχαμε περισσότερους πόρους θα μπορούσαμε να έχουμε στάξει μια μεγαλύτερη έκθεση και να καλύψουμε όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε. Δεν υπάρχει πλήρες κείμενο που να καλύπτει όλα τα σημεία που εσείς θέσατε. Νομίζω ότι εκφεύγουν του πεδίου αυτή τη έκθεση αυτά που θα σας ενδιέφεραν εσάς. Αυτά μπορώ να σας πω. Ωραία. Τώρα να ακούσουμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις και μετά θα δούμε αν υπάρχει χρόνος για απαντήσεις κατά την ε, παρούσα συνεδρίαση. Κυρία Μάκιντσα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Πρώτον, Ο αρμόδιος της ομάδας μου που εξέτασε το θέμα αυτό, δυστυχώς δεν ε, είναι σήμερα εδώ, είναι η Όλγα Στίβενς. Ήθελε να θέσει το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Πλούρα για μεταφράσεις. Θέλουμε και τις μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες. Μένα τα αγγλικά μου αρκούν, αλλά άλλα μέλη της ομάδας μου αυτή ήταν ε, η πρώτη ερώτηση. Επίσης θα ήθελε γιατί, να ήθελε να ρωτήσει γιατί αναφέρονται μόνο τρεις εμπειρογνώμονες όλη την έκθεση. Υπάρχει λόγος, είπατε ότι υπήρχαν έξι εμπειρογνώμονες. Αναφερθήκατε όμως μόνο τελικά σε εμπειρογνώμονες από την Ουγγαρία, τη Γερμανία και το Βέλγιο. Δεν ξέρω γιατί είναι αυτό. Επόμενη ερώτηση. Υπάρχει λόγος γιατί η παγκόσμια έκθεση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες του 2011 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που περιέχει τη γνώμη 370 εμπειρογνωμόνων. Γιατί δεν αξιοποιήθηκε για την έκθεσή σας εφόσον υπάρχει συγκεκριμένο κεφάλαιο για το κόστος των αναπηριών. Και τέλος, θεωρεί ότι δεν γίνονται επαρκές αναφορές στην αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για αυτό, η οποία λέγεται CRPD. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εξέφρασε ευχαριστίες για την εργασία σας. Να κάνω τώρα και μία ερώτηση δική μου. Είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακούσατε τα σχόλια του συναδέλφου Χάουιτ, που είναι επίσης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε μερικά καταπληκτικά υποδείγματα που πολύ θα ήθελα να έχετε κοιτάξει για το πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό. Αναφερθήκατε σε ένα προστατευμένο εργαστήριο συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Εγώ εργαζόμουν, έχω εργαστεί, έχω συνεργαστεί με μια οργάνωση που λέγεται Βασιλική Βρετανική Λεγεώνα για τις ε, βιομηχανίες. Δίνουν θέσεις εργασίας σε βετεράνους των ενόπλων δυνάμεων που έχουν ε, προβλήματα αναπηρίας ή προβλήματα πνευματικής υγείας οι μέθοδοι τους βεβαίως είναι μέθοδοι κοινωνικής απασχόλησης δίνουν όμως δυνατότητα απασχόλησης σε άτομα με ειδικέ ανάγκες και έχουν θαυμάσιο ποσοστό επιτυχίας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν τα κοιτάξατε αυτά και αν θα είχατε σχόλια. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέλιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την ε, ομάδα που μας παρουσίασε την έκθεση. Όλοι εκτιμήσαμε την έκθεση αυτή. Θέλω να διευκρινίσω κάτι από την πλευρά των επιχειρήσεων. Γιατί εγώ προέρχομαι από την επιχειρηματικό κόσμο. Παρά λοιπόν τα ωραία λόγια που ακούγονται στην ε, Ιταλία που είναι η χώρα που γνωρίζω καλύτερα ξέρω ότι για τις επιχειρήσεις ε, η χορήγηση εργασίας ε, στα άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρείται βάρος τις περισσότερες φορές και πολύ συχνά δημιουργείται η εντύπωση ότι η προσπάθεια που κάνουν για να βοηθήσουν ε, τα άτομα αυτά ε, δεν είναι προσπάθεια που γίνεται από όλη την κοινωνία, είναι προσπάθεια που επιβαρύνει μόνο τις επιχειρήσεις. Βεβαίως έχουμε κάνει αρκετά στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αλλά δεν έχουμε κάνει αρκετά στα πλαίσια της κοινωνίας γενικότερα. Δεν κάναμε την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει η νοοτροπία στην κοινωνία ευρύτερα. Αυτό το αποδεικνύουν και τα στοιχεία που αναφέρατε. Είπατε ότι παρά τις διάφορες πολιτικές το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα με ειδικέ ανάγκε, δυστυχώ είναι διπλό ε, σε σχέση με τον υπόλοιπο εργαζόμενο πληθυσμό και στην Ιταλία ιδιαίτερα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δυσχερής για τα αμαία ε, βέβαια δεν εξετάσετε την κατάσταση της Ιταλίας αλλά να έχετε υπόψη σας ότι έχουμε 680.000 ε, άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι γεγραμμένα στο σχετικό μητρό και τα τελευταία χρόνια μόνο 18.000 αμαία βρήκαν δουλειά. Ενώ θα έπρεπε ε, με βάση τις προβλέψεις μας να έχουμε βρει για 41.000 αμαία θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δεν πρέπει να είναι μόνο θεωρητικές οι δεσμεύσεις μας μέσω κανόνων δηλαδή, να υπάρξει πραγματική προσπάθεια στην κοινωνία, να αλλάξει η αντίληψη για τα αμαία. Το να θεωρείτε ότι είναι κόστος ε, η δουλειά που δίνουμε στα αμαία είναι εντελώ λάθος προσέγγιση. Δεν μπορούμε να αποστικοποιήσουμε πάντα, αλλά είναι βελτίωση της ποιότητας ζωής για τα αμαία. Είναι κάτι που δεν είναι απτό. Δεν μπορούμε να το εκφράσουμε σε ευρώ. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχουν κοινοί ορισμοί, συγκρίσιμοι ορισμοί για να είναι συγκρίσιμα και τα αποτελέσματα της έρευνας. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε πρότυπο. Σήμερα η κοινωνία αντιμετωπίζει τα αμαία ως μειονεκτούντα άτομα και θεωρείται ότι τα αμαία πρέπει να προσαρμοστούν στην κοινωνία. Αντίθετα, η κοινωνία πρέπει να προσαρμοστεί στα αμαία. Αυτή πρέπει να είναι η προσέγγιση. Επίσης, πρέπει να τονίσω ότι πρόσφατα υπόθηκε ότι είπε ο Υπουργός Εργασίας ότι δεν θα ανανεωθεί χρηματοδότηση για το ειδικό ταμείο για το 2015 για τα ΑΜΕΑ. Να, μία ακόμη καταστροφική είδηση, αν αυτό ε, επιβεβαιωθεί. Μέχρι τώρα λάβαναν λοιπόν κάποια επιδότηση, κάποια χρηματική ενίσχυση οι επιχειρήσεις που έδιναν εργασία στα ΑΜΕΑ. Αν τώρα καταργηθεί και αυτή η επιδότηση, δεν καταλαβαίνω τι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε. Πρέπει να δεσμευτεί και η αρμόδια επίτροπος, πρέπει να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα αμαία. Πρέπει να δεσμευθούμε, να αφιερώσουμε περισσότερες προσπάθειες για να μην ε, αντιμετωπίζουμε με τέτοιο τρόπο τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση, αλλά κατά την άποψή μας είναι σκανδαλώδης η αντιμετώπιση από διάφορες ε, οπτικές γωνίες. Βεβαίως ε, δεν ε, έχει κάποιο κόστος η βοήθεια προς τα αμαία, αλλά στην ουσία είναι ανεκτήμητη. Οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να βοηθήσει τα αμαία να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, πρέπει να θεωρείται θεμελιώδες εθνικό καθήκον και να χρηματοδοτείται πλήρως από το κράτος. Δεν μπορούμε καν να αντιμετωπίσουμε το θέμα της απόδοσης, της επένδυσης. Δεν υπάρχει καμία τέτοια αντίληψη. Να θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε αντιλήψεις παρόμοιες για όλους, συγκρίσιμες για όλους. Συγκρίνει τα αμαία με άτομα που δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα και αυτό είναι σκανδαλώδες. Αντίθετα, βεβαίως πρέπει να διαχειριζόμεθα καλύτερα ε, τα ποσά που πρέπει να διατίθενται για να βοηθάμε τα με αυτό είναι απαραίτητο. Μας ε, προτάθηκαν ε, διάφοροι προσανατολισμοί, ενδιαφέροντες όλοι αυτοί, αξιοποιήσιμοι σίγουρα και κυρίως συμπληρωματικοί. Θέλουμε να επιμείνουμε ιδιαίτερα και νομίζω ότι η έκθεσή σας όταν θα έχουμε δυνατότητα να τη διαβάσουμε πλήρως θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι σε όλες τις χώρες πρέπει να γενικευθεί η δημιουργία κέντρων της ε, βοήθειας μέσω της εργασίας. Εσείς τα λέτε προστατευμένους τόπους εργασίας. Έτσι θα βοηθήσουμε τα άτομα που έχουν ε, βαριές αναπηρίες που δεν μπορούν να βοηθηθούν σε συνήθεις τόπους εργασίας για ελαφρότερες αναπηρίες. Αν έχουμε τέτοια ειδικά κέντρα θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μόνιμες θέσεις εργασίας για τις βαρύτερες περιπτώσεις αλλά κυρίως θέσεις εργασίας προσωρινές για προσωρινές αναπηρίες μπορούν να λειτουργήσουν, μπορούμε να αποτιμήσουμε τη λειτουργία τους ευκολότερα και θα μας επέτρεπαν να αποτιμήσουμε και ακριβώς τι μισθούς πρέπει να δίνουμε και να δούμε και τι βοήθεια πρέπει να δώσουν ε, τα κράτη-μέλη για τις κοινωνικές κρατήσεις. Λοιπόν, εάν από την άλλη μεριά επιδιώξουμε πολύ βαριές κυρώσεις και ποσοστώσεις, πρώτα απ' όλα αυτά θίγουν την αξιοπρέπεια των ΑΜΕΑ αλλά ασκούν πίεση και στον κόσμο της εργασίας. Άρα δεν ανταποκρίνονται καθόλου ε, στην άποψη που έχουμε για την ε, κρατική κυριαρχία για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ, αλλά θα θέλαμε να έχουμε το σύνολο της έκθεσής σας σε κάθε γλώσσα. Αλλά επιμένω, τα κέντρα βοήθειας μέσω της εργασίας που εσείς τα αποκαλείτε προστατευόμενους τόπους εργασίας πρέπει να γενικευθούν θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε και τις επιπτώσεις της κρίσης γιατί αυτά τα κέντρα δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από τις οικονομικές κρίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στάινρουκ. Ναι, καταρχάς, κάτι άσχετο με την συζήτηση αυτή. Ε, χειμωνιάζει και κάνει κρύο στις αίθουσες. Πάλι θα πρέπει να βάζουμε τα παλτά μας για να καθόμαστε εδώ πέρα. Σας παρακαλώ, για πείτε το στους αρμόδιους, γιατί είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ τώρα για τις αναλύσεις σας, για τα έγγραφα, την μελέτη, πάρα πολύ εμπεριστατωμένα πορίσματα και θα πρέπει να τα μελετήσουμε. Σκοπός θα πρέπει να είναι ε, τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζουν μια ζωή με αυτοδιάθεση, χωρίς ε, εμπόδια σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Να επενθυμίσω ότι δεν είναι μόνο οι αναπηρίες εκγενετής που υπάρχουν. Ανά πάσα στιγμή στον καθένα μας μπορεί να τύχει το οτιδήποτε. Και την πολυμορφία των αναπηριών που υπάρχουν. Αν σωστά κατάλαβα, και αυτή είναι η ερώτησή μου, είναι σημαντικό στην Ευρώπη να κινηθούμε προς την κατεύθυνση κοινών ορισμών. Να δούμε τι μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση και ποια θα μπορούσαν να είναι τα ελάχιστα κοινά πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι επίσημη αναγνώριση των αναπηριών. Για το θέμα των ποσοστώσεων τώρα. Από τη Γερμανία είμαι και ξέρω το σύστημα των ποσοστώσεων πάρα πολύ καλά. Σωστά κατάλαβα. Μιλάτε για μεγάλα πλεονεκτήματα για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία και ότι οι κυρώσεις μέσω των ποσοστώσεων όταν χρησιμοποιούνται στοχευμένα, μπορούν να υποστηρίξουν την κοινωνία σε ό,τι αφορά την κατάργηση των εμποδιών, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η νόμοι τώρα για την κατάργηση των εμποδίων είναι πάρα πολύ σημαντική σε κάθε περίπτωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα εργασίας της το 2014 σκόπευε να υποβάλει μια τέτοια πρόταση. Δεν το έχει πράξει ως τώρα. Εγώ είμαι από την Ινανία Βεσφαλία στη Γερμανία και έχουμε από το 2003 νόμο για την υποχρέωση κατάρχηση των εμποδίων πρόσβασης. Είναι πολύ καλό το νομοσχέδιο. Ήταν πολύ καλός ο νόμος, εύκολο στην εφαρμογή του. Κάτι άλλο που δεν άκουσα στην ανάλυση σας, αλλά δεν ήταν και στην ε, εντολή σας. Έχουμε μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά με συγκεκριμένες ελευθερίες. Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσον τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτή την ενιαία εσωτερική αγορά. Πριν από κάποιες ημέρες ήμουν με μια ομάδα ατόμων με διάφορες αναπηρίες και με φρίκη άκουσα ότι ο εθνικός ε, βοηθός ε, στην Γερμανία δεν μπορεί να περάσει τα σύνορα προς τη Γαλλία. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Δηλαδή, αν θέλει κανείς από το κρατήδιό μου να πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν μπορεί να έχει τον βοηθό του μαζί. Πιστεύετε ότι υπάρχει λοιπόν ανάγκη να δώσουμε πιο πολύ ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο πολύ Ευρώπη στα άτομα με αναπηρία. Και τελευταία ερώτηση. Ε, έχετε ασχοληθεί για το κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μία ταυτότητα για αμαία. Και ποιο θα ήταν και το όφελος, μιας και όλα αυτά ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο με πολύ διαφορετικό τρόπο. Έχουμε ευρωπαϊκά συμβουλία εργαζομένων. Έχουμε ευρωπαϊκές εταιρείες που ασχολούνται με τα άτομα με αναπηρία. Θα είχε νόημα να ζητήσουμε βελτίωση των όρων, των συνθήκων, να δημιουργήσουμε για παράδειγμα ευρωπαϊκά συμβούλια εργασίας. Ο κύριος Φουντούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εξετάσαμε σύμφωνα με τη μελέτη το ισοζύγιο μεταξύ κόστους και απόδοσης των επενδύσεων για λελογισμένες προσαρμογές όσον αναφορά τα αμαία. Δηλαδή, εάν αξίζει να επενδύσουμε από οικονομικής πλευράς στο δικαίωμα στην εργασία των ατόμων με αναπηρίες. Αυτό που δεν μπορεί να μετρηθεί με χρήματα και είναι πολύ σημαντικό είναι το κοινωνικό όφελος. Τα άτομα με αναπηρίες που βρίσκουν μια θέση εργασίας αισθάνονται ότι προσφέρουν και η χαρά που λαμβάνουν όταν αμείβονται δεν μπορεί να μετρηθεί με χρήματα. Σαν πατέρα μια κόρη 30 ετών με σύνδρομο Down και έχω ασχοληθεί ενεργά με το θέμα τη ένταξη στην αγορά εργασία των ατόμων με αναπηρία, χαίρομαι γιατί η μελέτη σχετικά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά το θέμα τη επιδότηση των θέσεων εργασία πρέπει να γίνεται με λελογισμένα και με πολύ προσοχή γιατί τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να αισθάνονται ότι τους δίνεται ευκαιρία για εργασία από Μην ξεχνάμε ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει αμαία. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι δεδομένο. Ένα ατύχημα στη ζωή μας και όλα μπορούν να ανατραπούν. Ας συνεχίσουμε λοιπόν προς αυτή τη θετική κατεύθυνση. Επίσης θα ήθελα να είχαμε τη μελέτη και στις άλλες γλώσσες για να μπορέσουμε να τη ε, μελετήσουμε ευκολότερα και αναλυτικότερα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τις ε, παρεμβάσεις σας, για τις ερωτήσεις που κάνατε. Σε ό,τι αφορά το πρακτικό σκέλος, θα γίνει συζήτηση με το τμήμα χαραξής πολιτικής και ίσως αυτό θα πρέπει να το συζητήσουν και οι συντονιστές. το κόστος για τις ε, διάφορες γλώσσες και η δυνατότητα χρηματοδότησης. Τα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν θα απαντηθούν γραπτά. Θα λάβετε γραπτές, σύντομες απαντήσεις από τους υπεύθυνου. Εν συντομία, λοιπόν, θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά γραπτά και με άλλους τρόπους. Είμαι βέβαιη ότι στη διάρκεια της θητείας αυτής το θέμα και η συζήτηση θα επανέλθει με διάφορες μορφές στη συζήτησή μας και στην ημερήσια διαταξή μας. Σας ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη νέες μορφές εργασιακών σχέσεων. Θα μας το παρουσιάσει η Eurofound. για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, συμπεριλαμβανομένης και της Νορβηγίας, σε ό,τι αφορά τις νέες μορφές απασχόλησης. Θα μας ε, κάνουν λοιπόν την παρουσίασή τους και ελπίζουμε να έχουμε το χρόνο να κάνουμε κάποια σχόλια πριν ε, ολοκληρωθεί ο χρόνος που προβλέπεται για την συνεδρίασή μας. Να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ειρήν Μάντλ, η οποία είναι υπεύθυνη από το Eurofound. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε κάποια από τα πορίσματά μας για τις νέες μορφές απασχόλησης και σχέσεις εργασίας. Πριν από δύο εβδομάδες σας ενημέρωσε ο διευθυντής μας ότι ε, ο ρόλος του Eurofund ε, δίνει πληροφορίες σε διάφορους τομείς ε, που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και φυσικά η απασχόληση είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα που μας απασχολούν, ξεκινήσαμε ένα νέο πρόγραμμα έρευνας για τις νέες μορφές εργασίας, διότι βρήκαμε ε, ε, κάποια στοιχεία, τεκμήρια και έγιναν και συζητήσεις για αυτές τις νέες μορφές εργασίας και μας δημιουργήθηκε η εντύπωση δεν είναι ξεκάθαρο ποιες είναι αυτές οι νέες μορφές εργασίας, ε, ποια, ποια, είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των αναδειωμένων μορφών εργασίας εργασίας και πώς επηρεάζεται η αγορά εργασίας από αυτές. Αυτό ήταν ο στόχος ε, του, ε, της μελέτης που κάναμε ε, για να κάνουμε και κάποιες συστάσεις για την εκπόνηση πολιτικής. Τι εννοούμε λοιπόν με νέα μορφά εργασίας. Ε, φαντάζεστε ότι είναι ετερογενείς αυτές οι μορφές εργασίας ε, λόγω των διαφορετικών μορφών εργασίας, των διαφορετικών νομοθεσιών που ισχύουν, διαφορετικών ε, παραδόσεων ως προς τις συλλογικέ συμβάσεις εργασίας και τον κοινωνικό διάλογο. Όλες οι μορφές εργασίας λοιπόν διαφέρουν. υιοθετήσαμε μια εθνική προσέγγιση και ζητήσαμε τους εθνικούς εμπειρογνωμούς να μας πούν δουν τι ε, καινούριο υπάρχει σε εθνικό επίπεδο, τι καινούριο συνάντησαν σε σχέση με αυτά που προϋπήρχαν για τη σχέση εργασίας, ε, δηλαδή ποια σχέση έχει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο ε, απομακρυνόμενη από το ένας προς έναν. Ένας εργοδότης, ένας εργαζόμενος. Μπορεί ένας εργοδότης να προσλάβει μια ομάδα εργαζομένων, μια ομάδα εργαζομένων να βρουν έναν, έναν εργοδότη ε, ε, επίσης σε διαφορετικά μοντέλα εργασίας, ε, δηλαδή παραδοσιακά έχετε ένα σετ καθηκόντων μέσα σε μια σύμβαση ορισμένου χρόνου και πέρα από την εξαρτημένη εργασία τώρα και όχι μόνο για τους αυτοαπασχολούμενους αποφασίσαμε να εξετάσουμε τις νέες μορφές συνεργασίας, ε, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες που λειτουργούν με συμβάσεις έργων. από το 2000 και μετά αρχίσαμε να εξετάζουμε την κατάσταση. Νέες νομοθεσίες, νέες συλλογικέ συμβάσεις εργασίας, νέες πρακτικές στις επιχειρήσεις, νέα νομοθετικά πλαίσια. Όλα αυτά μελετήσαμε είναι οι νέες μορφές εργασίας. Ε, βάσει της ε, μελέτης μας αλλάζει, όπως είπαμε, η σχέση εργασίας. Στη συνέχεια υπάρχουν και διαφορετικές ε, ε, διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης ε, της εργασίας. Ε, φυσικά υπήρχαν επικαλύψεις ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα και στο κάτω μέρος της λίστας ασχολούμαστε με τους αυτοαπασχολούμενους και τις νέες μορφές συνεργασίας. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, δεν θα μου δοθεί η ευκαιρία να σχολιάσω και τις εννέα αυτές αναδυόμενες μορφές εργασίας. Θα επικεντρωθώ σε κάποιες για να σας δώσω κάποιε κάποιες λεπτομέρειες. βλέπετε με κόκκινο τις νέες μορφές που θα σχολιάσω. Employee sharing, επιμερισμό επιμερισμός εργαζομένων δεν προσλαμβάνει ένας εργοδότης έναν εργοζόμενο, αλλά γίνεται με ομάδες. Δηλαδή υπάρχει μια ανεξάρτητη οντότητα που λειτουργεί ως εργοδότης και αυτή η οντότητα στέλνει τον εργαζόμενο στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, όπως λίγο γίνεται με τις, ε, με τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, όμως ε, δεν ξέρουμε εκ των προτέρων σε ποιες επιχειρήσεις θα πάει ο εργαζόμενος, γιατί λειτουργεί αυτό μόνο με ε, εταιρείε μέλη. Έχει μια περιφερειακή διάσταση. Α, και δεν χρειάζεται να είναι επιχείρηση. Μπορεί να είναι και δημόσιο φορέα ή με κρατικό φορέα. Ε, ε, υπάρχει η ευθύνη για του εργαζόμενου. Δεν αγοράζουν, δεν νοικιάζουν εργαζόμενου, αλλά ε, έχουν την ευθύνη για την εργασία που του αναθέτουν. Και η νομική οντότητα που συστήνεται για να λειτουργήσει ω εργοδότη για αυτούς τους εργαζομένους ε, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Φυσικά θα αποκομίσει κάποιο κέρδος, αλλά βασικό στόχος είναι να παράσχει πλήρη απασχόληση στους εργαζομένους ε, συνδυάζοντας ε, ανάγκες ανθρωπίνων πόρων διαφόρων επιχειρήσεων που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν μερική απασχόληση. Αυτό σημαίνει πως για τον εργαζόμενο είναι θετικά, θετικά τα αποτελέσματα ή ενδυνάμει θετικά και για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες, ε, διότι για τους εργοδότες υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό παρότι δεν μπορούν να προσφέρουν πλήρη απασχόληση και για τους εργαζομένους ε, προσφέρει σταθερή απασχόληση διότι στις περισσότερες περιπτώσεις ε, είναι πλήρης απασχόληση μόνιμη και, καλύπτεται αυτό το κενό όταν δεν υπήρχε νωρίτερα δηλαδή αρκετή ζήτηση για αυτή τη δουλειά. Είναι win-win, ε, αμοιβαίως επικερδής η κατάσταση και για τους εργοδότες και για τους εργαζομένους και, χάρη στην περιφερειακή διάσταση αυξάνεται η ελκυστικότητα των περιφερειών, ε, σταθερότερη απασχόληση, εξειδικεμένο προσαπικό που ε, χρειάζεται πλέον σε εκείνη την περιοχή λόγω της ομαδοποίησης. Δεύτερη μορφή εργασίας, casual work, ε, εκπεριτροπής εργασία ή ε, περιστασιακή εργασία ε, με διαλύματα ή η εργασία σε επιφυλακή. Τι σημαίνει σε επιφυλακή. Ε, μία μονιμότερη σχέση εργασίας, αλλά ο εργοδότης ε, δεν υποχρεούται να δίνει δουλειά στον εργαζόμενο, όχι καλεί τον εργαζόμενο όταν τον χρειάζεται. Ο εργοδότης λοιπόν ε, έχει μεγαλύτερη, διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία και Ορισμένες φορές όμως είναι υπερβολική ευελιξία, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα προγραμματισμού, σχεδιασμού και σταθερότητας, ε, διότι ποικίλει ο τρόπος ε, που του ε, καλεί ο εργοδότης, ε, ορισμένες φορές είναι πάρα πολύ βραχυπρόθεσμα, τους παίρνουν σήμερα το πρωί για να έρθουν για δύο ώρε. παραδείγματο χάρη, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος και άρα ε, υπάρχει αστάθεια για τον εργαζόμενο. Θεωρητικά μπορούν να, όταν λαμβάνουν την κλίση, να απορρίψουν την προσφορά του εργοδότη. Εάν βεβαίω το κάνουν αυτό υπερβολικά συχνά, δεν του ξαναπέρνουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι περιορίζεται το περιθώριο ελιγμών τους για την ασφαλιστική προστασία, την κοινωνική ασφάλιση θεωρητικά και πάλι εδώ φαίνονται πολύ ωραία αυτά διότι είναι μόνιμες οι συμβάσεις ε, οπότε ε, δικαιούνται και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όμως στην πράξη μπορεί να τους καλούν συχνά ή όχι και ανάλογα με τη συχνότητα να μην δικαιούνται τις ασφαλιστικές παροχές γιατί τα περισσότερα εθνικά συστήματα αυτά είναι συνάρτηση των ωρών ή ημερών που έχει αποσχοληθεί ε, κάποιος για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους αυτό το τύπο εργασίας έχουμε και άλλα χαρακτηριστικά παρατηρείται μεγαλύτερη ζήτηση σε τομείς όπου υπάρχουν μεγάλες διακοιμάνσεις ή έχουν ιδιαίτερα εποχιακό χαρακτήρα ε, οι θέσεις και έτσι καλύπτονται μεγάλα κενά ανθρωπίνων πόρων. Είναι χαμηλής η ε, θέση εργασίας και κυρίως ε, απευθύνονται σε γυναίκες. Υπάρχει ένα είδος εδώ ε, κατάτμησης, κατακαιρματισμού της αγοράς εργασίας και βασιζόμαστε την ε, ζήτηση από πλευράς εργοδότη αλλά από πλευράς ε, εργαζομένου δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση. Το κάνουν διότι δεν έχουν καλύτερη εναλλακτική λύση, επειδή τους αρέσει. Ε, για τις ε, επιπτώσεις ε, για την αγορά εργασίας και για τις συνθήκες εργασίας βλέπετε ότι είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση σε σχέση με την πρώτη διαφάνεια, δηλαδή πολύ περισσότερες ενδυνάμει αρνητικές επιπτώσεις κατά τη διαστολή με τις θετικές και είναι μάλλον επισφαλής η θέση του εργαζομένου. Μια άλλη νέα μορφή είναι η κινητή εργασία που βασίζεται στις ε, τεχνολογίες ε, πληροφορίας ε, εκτός χώρου εργασίας του πελάτη, εξ αποστάσεως, όπως το... Δεν ασχολούμαστε με την παραδοσιακή τηλεεργασία, αλλά εξετάζουμε πιο κινητές μορφές εργασίας. Αυτό σημαίνει πως και πάλι είναι εξαιρετικά ευέλικτη αυτή η μέθοδος εργασίας, αλλά ε, κατά τη διαστολή με τη τηλεεργασία οι εργαζόμενοι ε, προσφέρουν την εργασία τους, όμως εδώ αντίθετα με την σε εργασία είναι πολύ εξειδικευμένο το προσωπικό και διατίθεται να ε, λειτουργήσουμε αυτόν τον ε, τρόπο που ε, βασίζεται στη μεγάλη κινητικότητα και στη χρήση νέων εργαλείων, υπολογιστές, iPads, FEE, τηλέφωνα κτλ. Υπάρχουν οι θετικές πτυχές γιατί όπως είπαμε προσφέρουν στον εργαζόμενο την ευελιξία που επιθυμεί προσφέρουν αυτονομία, καλύτερη δυνατότητα οργάνωσης ε, της εργασίας και άρα μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη παραγωγικότητας, ε, κάτι που δύσκολα επιτυγχάνεται σε ένα παραδοσιακό χώρο εργασίας όπου κανείς υποχρεούται ε, να υπαχθεί σε αυτό το πατριαρχικό σύστημα οργάνωσης εργασίας, δηλαδή επιβάλλει εργοδότη τον τρόπο εργασίας. Από την άλλη, Υπάρχουν αρνητικές επιτυχές. 24 ώρες το 24ωρο πρέπει να είναι διαθέσιμος ο εργαζόμενος και άρα έχει μεγαλύτερο άγχος και πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Κοινωνική απομόνωση επίσης, διότι ε, μπορεί να, πηγαίνουν, να δουλεύουν οπουδήποτε, αλλά να μην έχουν σχέση με τον κοινωνικό ιστό. Η, νέα μορφή, α, μια, η επόμενη μορφή εργασίας ε, σχετίζεται με τις επιταγές εργασίας. Ε, ε, είναι μια επιταγή που χρησιμοποιεί ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε περισσότερες περιπτώσεις ένας δημόσιος φορέας προσφέρει αυτά τα κουπόνια και τα κουπόνια καλύπτουν όχι μόνο το μισθό, αλλά και ένα μέρος ε, της ε, κοινωνικής ε, προστασίας, σε περισσότερες περιπτώσεις κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος. Ο βασικότερος λόγος θέσπιση ενό τέτοιου συστήματο, όπω είδαμε στι χώρε που το έχουν, είναι να νομιμοποιήσουν την εργασία κυρίω στον τομέα τη γεωργία και των κατοίκων υπηρεσιών. Στην πράξη, αυτό διαπιστώσαμε, αυτή είναι η βασική τομή και σε κάποιες χώρες έχουν εισαχθεί και περιορισμοί ε, ως προς τους εργαζόμενους εργοδότες ή το πεδίο που μπορεί να καλυφθεί με αυτά τα κουπόνια. Ε, ο στόχος και πάλι είναι να μην εκτοπιστούν άλλες ε, μορφές εργασίας νομιμοποιώντας αυτή. Οι επιπτώσεις είναι μικτές και πάλι, έχουμε αρνητικά και θετικά ευρίσματα. Ε, νομιμοποίηση της ε, μη δηλωμένης εργασίας. Ο εργαζόμενος ε, επίσης έχει κοινωνική προστασία, αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Από την άλλη υπάρχουν και αρνητικέ επιτυχίες και πάλι κοινωνική απομόνωση, κυρίως για τις κατοίκων υπηρεσίες, διότι τι σημαίνει αυτό ότι η οικογένεια λείπει, έχουν πάει στη δουλειά, στο σχολείο και κάθονται μόνοι τους μέσα στο σπίτι και δουλεύουν, δεν έχουν σε επαφή με κανέναν. Ε, συμπεράσματα και κάποιες συστάσεις για την ε, πολιτική. Ε, βασική κινητήριο σε δύναμη για τις νέες μορφές εργασίας, όπως θα διαπιστώσατε, είναι η ευελιξία που ζητάει είτε ο εργοδότης, είτε ο εργαζόμενος, είτε και οι δύο είδαμε ότι κάποιες ε, μορφές απασχόλησης έχουν ε, ε, κάποιο δυναμικό διότι είναι αμοιβαίως ε, επικερδείς, άλλες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, όπως η σε εργασία, κυρίως στις κινητές θέσεις εργασίας ε, ICT, στον τομέα της πληροφορικής. Δεν σας μίλησα καθόλου για το crowd employment, ε, άλλη μια νέα μορφή εργασίας, αλλά υπάρχουν αρνητικές επιτυχίες Κάτι άλλο. Ε, σε αυτές τις νέε μορφές που εντοπίσαμε υπάρχουν εγγενή καλά χαρακτηριστικά ε, και μπορούν να οδηγήσουν σε διαρθρωτικού τύπου αλλαγές στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κυρίως για το χώρο εργασίας. Απομάκρυνση από το χώρο στον οποίο βρίσκεται ο εργοδότης. Επίσης, επιρροή επί των ωραρίων εργασίας, κατακαιρματισμός ή πιο ανεξέλεγκτα ή μη ελέγξιμα ωράρια εργασίας για τα μοντέλα εργασίας ε, μπορεί πλέον, να μην μιλάει για δουλειά αλλά για καθήκοντα, έργο, για έργα ε, που πρέπει να επιτελεστούν περιορισμένης ε, εμβέλειας. Τώρα, εάν χρειάζεται παρέμβαση από πλευράς αυτών που εκπονούν την πολιτική σε μακροοικονομικό επίπεδο θα λέγαμε για κάποιες μορφές εργασίας όχι, διότι είναι, έχουν, αντιστοιχούν στην ε, ε, μειοψηφία των θέσεων στην αγορά εργασίας και συνδέονται με το ε, κάποιο είδος εργοδοτών εργαζομένων ή καθηκόντων. Ε, ή με συγκεκριμένου τομεί. Ε, σε άλλε πάλι περιπτώσει θεωρήσαμε ότι χρειάζεται παρέμβαση, κυρίω για τι μορφέ εργασία που ενδυνάμει έχουν ε, πολλά προνόμια για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους διαπιστώσαμε ότι στην αγορά εργασίας δεν υπάρχει μεγάλη συνειδητοποίηση, ευαισθητοποίηση ότι υπάρχουν αυτές οι μορφές εργασία μπορούν να προσφέρουν πολλά, ίσως θα έπρεπε να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση και με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε μεγαλύτερα ωφέλη και να έχουμε κάποια κίνητρα για να ενθαρρύνουμε αυτές τις μορφές εις βάρος άλλων που είναι αρνητικές. Ε, επίσης για τις αρνητικές μορφές εργασίας δεν χρειάζεται απαραίτητα νομικό πλαίσιο. Ίσως ε, συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή ε, κώδικες σε προαιρετική βάση θα μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο ώστε να έχουμε ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων από τις ενδυνάμει αρνητικές επιπτώσεις. Τέλος, επειδή είδατε ε, ότι είναι ετερογενής οι μορφές εργασίας ε, θα προτείναμε αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει για τον τρόπο με τον οποίο ε, μπορούν να σχεδιαστούν οι μελλοντικές εξελίξεις για τις νέες μορφές εργασίας για να είναι κατά το μέγιστο ε, επικερδής για όλους. Αυτά ήθελα να σας πω και με τα χαρές να απαντήσω και σε όποιες ερωτήσεις υπάρχουν. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ε, λίγα λεπτά έχουμε αν υπάρχουν ερωτήσεις ε, που θέλετε να κάνετε στην κυρία Μάντεν πριν ε, χρειαστεί να φύγει για την Ιρλανδία. Παρακαλώ, έχετε ερωτήσεις η κυρία Στάνιοκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας, για την παρουσίασή σας. Είναι πολύ σημαντικό ο μεταβαλλόμενος τρόπος εργασίας, τόπος εργασίας, να παρατηρηθεί. Πολλές αλλαγές γίνονται για λόγους εισαγωγής ε, τεχνολογιών και είναι θετικές, αλλά ορισμένες ε, σύγχρονες ε, μορφές απασχόλησης σίγουρα πρέπει να μας απασχολήσουν. Πρέπει να προσέξουμε ότι η ευελιξία για τις επιχειρήσεις να έχει κάποια σύνορα. Να μην εμποδίζει τους εργαζόμενους να τα βγάζουν πέρα. Όταν βλέπω αυτά τα συνεχόμενα συμβόλαια όπου πρέπει να είναι κανείς σε επιφυλακή χωρίς ποτέ να ξέρει αν θα απασχοληθεί και θα αμυφθεί τότε πιστεύω ότι πρέπει να παρέμβουμε για να δούμε εάν η νομοθεσία η ευρωπαϊκή και η εθνική είναι επαρκής για να αντιμετωπίσει όλες αυτές ε, τις μορφές εργασίας. Έχουμε την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Αλλά πρέπει να δούμε πώς ε, λαμβάνει υπόψη αυτούς τους χρόνους επιφυλακής και τι όρια θέτει. Από ό,τι κατάλαβα προτείνεται και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν μια διαρθρωμένη ανταλλαγή απόψεων για αυτές τις μορφές εργασίας. Δεν ξέρω αυτά τα συμβόλαια στα οποία αναφερθήκατε υπήρχαν μόνο στο Ενωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα ορισμένες τέτοιες μορφές και στη Γερμανία. Έχω όμως την εντύπωση ότι διευρύνεται και σε άλλες χώρες η χρήση τους. Τώρα μια ερώτηση. Αυτή η εργασία ε, κατά τμήματα της ε, επιμεριζόμενης εργασίας λοιπόν πώς μπορούμε να την ε, προσαρμόσουμε τόσο ώστε να είναι θετική για όλους. Και επίσης αυτή η διακεκομένη εργασία επίσης ε, σε ποιο ε, νομικό πλαίσιο βασίζεται στις διάφορες ε, χώρες μέλη όπου υπάρχει και τι διαφορές υπάρχουν. Κατά πόσο αξιοποιείται και τι καθήκοντα έχουν οι εργαζόμενοι που εργάζονται με αυτόν τον τρόπο εργασίας. Ο κύριος Μπάχτου και μετά να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και την εργασία που επιτελέσατε. Νομίζω για την πολιτική μας εργασία είναι πολύ χρήσιμη. Δύο ερωτήσεις. Αναλύσατε τέσσερις νέες μορφές εργασίας. Έχετε επιπλέον πληροφόρηση για τους τομείς όπου χρησιμοποιείτε οικοδομές, μεταφορές, για παράδειγμα, πού χρησιμοποιούνται. Μιλήσατε για τις εποχιακές δραστηριότητες, για τη γεωργία, Μήπως έχετε πληροφορίες για τους τομείς όπου αξιοποιούνται, χρησιμοποιούνται αυτές οι νέες μορφές εργασίας. Η δεύτερη ερώτηση συνδέεται με αυτό που είπε και η κυρία Στάινρουκ. Θα ήταν σημαντικό να μας δώσετε επιπλέον πληροφόρηση γιατί συζητούμε τώρα την οδηγία πλαίσιο του 98 για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Θα μας βοηθούσε λοιπόν επιπλέον πληροφόρηση για τα σημεία που θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε σε αυτή τη συζήτηση και αυτή την οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας. Πρώτον, θεσμοθετημένη ανταλλαγή απόψεων. Ναι, αυτό προτείνουμε και στο εσωτερικό της κάθε χώρας για να εξετάσουμε καλύτερα την κατάσταση μεταξύ των διαφόρων ε, κλάδων, μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και γενικότερα μεταξύ των χωρών. Ορισμένες από αυτές τις μορφές ε, απασχόλησης είχαμε αυτήν, ξέρετε, την ε, αντιμετώπιση κατά κράτος. Είχαμε αυτή τη νέα μορφή job sharing, επιμορισμού της εργασίας Οι μορφές ε, αυτές είναι πολύ νέες σε κάποιες χώρες, αλλά όχι σε άλλες. Γι' αυτό θα προτείναμε μια πιο πανευρωπαϊκή ανταλλαγή απόψεων για το τι διδάγματα έχουμε εξαγάγει, τι πρακτικές έχουν εφαρμοστεί. Στα νέα κράτη-μέλη, για παράδειγμα, πρόσφατα υπήρξε νομική βάση για αυτή τη μορφή εργασίας. Από τις μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μεγάλη σύγχυση και μεταξύ εργοδοτών και μεταξύ εργαζομένων. Γιατί αυτή η νομική βάση ήταν τόσο περίπλοκη για να εγγυάται τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων που ήταν δυσνόητη. Άρα ε, ίσως η πείρα ε, των χωρών που έχουν αξιοποιήσει περισσότερο χρόνο αυτό τον τρόπο εργασίας ε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Δεν χρειάζεται κάθε φορά κάθε χώρα να επανεφευρίσκει τον τροχό. Ορισμένες ε, μορφές εργασίας ήταν τόσο νέες που εμείς ε, βρήκαμε όνομα για αυτές. Υπήρχαν διάφορες ε, παραλλαγές τους σε διάφορες περιοχές της χώρας αλλά δεν υπήρχε όνομα. Καλύτερα λοιπόν να επιδιώξουμε μια ευρωπαϊκή προσπάθεια ε, σύγκριση και ορισμού τους, ιδίως εκεί που έχουμε αρνητικές επιπτώσεις, για να τις μετριάσουμε. Αυτή τώρα η, ε, αυτός ο επιμερισμός εργαζομένων, πώς λειτουργεί στην πράξη. Στη Γερμανία και την Αυστρία λέγεται Arbeitgeber Zusammenschluss ή Group Mount στη Γαλλία και το Βέλγιο. Αυτές είναι οι έννοιες και παρόμοια έχουμε δει και στη Φιλανδία και την Ουγγαρία. Πώς λειτουργεί. Είναι πολύ περιφερειακό όργανο από στρατηγικής πλευράς. Δηλαδή, στις περισσότερες περιπτώσεις, κάποιος εμπλεκόμενος μπορεί να έχει θεσμικό χαρακτήρα ή να είναι κάποιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή να είναι μια εταιρεία που κάνει μια ανάλυση σε περιφερειακό επίπεδο, να δουν αν υπάρχει ζήτηση για να μοιράζονται κάποιοι εργοδότες, κάποιους εργαζόμενους. Και αν καταλήξουν ότι υπάρχει περιθώριο, έρχονται σε επαφή με τις εταιρείε να τις ρωτήσουν αν θέλουν να συμμετάσχουν και αν υπάρχει επαρκής μάζα και επιχειρήσεων και εργαζομένων αυτή η οργάνωση Αιγίδα δημιουργείται, αναλαμβάνει το κόστος ε, το διοικητικό, προσλαμβάνει, επιλέγει, είναι σαν παραδοσιακός εργαζόμενος από την διοικητική πλευρά και συντονίζουν με τις επιχειρήσεις ποιος χρειάζεται ποιον εργαζόμενο πότε. Έτσι αρχίζει να λειτουργεί. Αυτό μπορεί να γίνει. Οι εργαζόμενοι λοιπόν εργάζονται εκ, περιτροπής στις επιχειρήσεις και οι όροι της περιτροπής ποικίλουν. Μπορεί να αλλάζουν δύο φορές την ημέρα επιχείρηση ή αναεξάμεινο. Εξαρτάται από τον τύπο εργασίας και τη ζήτηση που υπάρχει. Είναι αναπερίπτωση λοιπόν, άρα πολύ ευέλικτο αυτός λοιπόν ο συντονιστικός φορέας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να είναι σε επαφή με όλους, πρέπει να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν και βεβαίως και αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι κάπως ευέλικτες. Αν μια επιχείρηση δεν μπορεί, ε, για παράδειγμα, να αξιοποιήσει τους εργαζομένους που είχε ζητήσει, να μπορεί να τους αναλάβει κάποια άλλη εταιρεία. Τώρα για την περιστασιακή ευκαιρική εργασία και τα κουπόνια. Υπάρχουν διάφορες ε, περιπτώσεις. Ε, έχουμε μιλήσει για τη διακεκομένη εργασία και τις ε, περιόδους επιφυλακής. Η διακεκομένη εργασία σε διάφορες χώρες, Βέλγιο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Σλοβενία, έχει νομικό πλαίσιο. Με διαφορετικά ονόματα, διαφορετικές λεπτομέρειες και για τις δύο αυτές μορφές σε ορισμένε περιπτώσεις αφορά μόνο κάποιους κλάδους. Σε άλλες υπάρχουν κανονισμοί για το πόσες ώρες, πόσες ημέρε μπορεί να εργαστεί ο κάθε εργαζόμενος ή πόσες μπορεί να παραγγείλει ένα εργοδότης. Παραδείγματα, στο Βέλγιο διαπιστώσαμε ότι στον τουριστικό κλάδο τα συμβόλαια είναι για δύο μέρες επειδή υπάρχουν μέγιστα ζήτησης και υπάρχει ο περιορισμός ότι κάθε εργοδότης μπορεί να αξιοποιήσει μόνο για 100 μέρες το χρόνο αυτούς τους περιστασιακά εργαζόμενους και κάθε εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί μόνο 50 μέρες ως περιστασιακά εργαζόμενος το χρόνο και επίσης δίδεται ένα καταποκοπήν ποσό για την κοινωνική ασφάλιση ανεξάρτητα λοιπόν από τι πληρώνει ο εργοδότης τον εργαζόμενο πρέπει να δώσει 7,5 ευρώ την ώρα σε Κοινωνικέ συνεισφορέ. Άλλο παράδειγμα στη Σλοβενία για να δοθεί δουλειά σε νέου και όπου μπορεί να δοθεί δουλειά μόνο σε νέου μεταξύ 15 και 26 και φοιτητέ. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. εντελώ διαφορετική προσέγγιση. Ο εργοδότη και ο εργαζόμενος δεν συνεργάζονται απευθεία. Υπάρχουν ειδικέ ε, εταιρείε, ε, οργανισμοί εξέφρασης εργασία για την επιφυλακή Είπατε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνεται πολύ. Δεν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη και δεσμευτική νομική βάση. Είναι δυνατό όμως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε άλλε χώρες, στην Ιταλία, την Ολλανδία, επίσης και μέρη στην Ιρλανδία, υπάρχει συγκεκριμένο κανονισμός για τα συμβόλαια αυτά επιφυλακή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τι πρόβλημα έχουμε. Ορισμένε φορέ δεν είναι σαφέ ποιο είναι το καθεστώ του εργαζόμενου είναι εργαζόμενος, είναι αυτοαπασχολούμενος, είναι υπάλληλο. Και μπορεί το καθεστώς ε, να αλλάζει όσο είναι σε επιφυλακή να είναι ένα και μόλις κληθεί να δουλέψει να είναι άλλο. Για τα κουπόνια υπάρχουν διαφορετικά συστήματα. Τέθηκε το ερώτημα σε ποιους τομείς. Είναι κυρίως στη Γεωργία, σε χώρες όπως η Λιθουανία, αλλά στις περισσότερες χώρες είναι κυρίως για εργαζόμενους ε, στο σπίτι, για οικιακούς και οικιακές βοηθούς. Βέλγιο, Αυστρία, επίσης για διάφορες ε, ε, εργασίες όπου βοηθάνε συγκεκριμένες εκδηλώσεις ή συγκεκριμένες διαφημιστικές εκστρατείες. Έχουμε δει διαφορετικά συστήματα. Ή υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενο, ενώ στο Βέλγιο και εν μέρη στη Γαλλία υπάρχει και ένας ενδιάμεσος οργανισμός που προσλαμβάνει τον εργαζόμενο με αορίστου ή ορισμένου πλήρους ή μερικής απασχόλησης υπάρχει αυτή η ευελιξία και ο ενδιάμεσος οργανισμός μετά στέλνει τον εργαζόμενο ε, για την ε, εργασία οικιακού βοηθού και ε, παίρνει ένα βάουτσερ ο εργαζόμενος, ε, ένα κουπόνι. Για την ευκαιριακή εργασία, αυτό κυρίως είναι εποχιακή, τουρισμός, ε, κατασκευές, γεωργία, αλλά και άλλοι τομείς όπου υπάρχει πολύ μεγάλη διακύμανση της ζήτησης. Και κάτι που είναι ιδιαίτερα ανισχυτικό είναι βεβαίως πολύ χαμηλόμιστες ενασχολήσεις και χαμηλού επίπεδου ειδίκευσης τομής. Ε, εδώ τα μοντέλα που έχουμε ε, είναι στη Γαλλία ε, τα συμβόλαια ξεκίνησαν από τη Γεωργία τώρα όμως ισχύει και σε άλλους τομείς και σε άλλες χώρες ισχύει σε πολλούς τομείς αλλά στην πράξη λειτουργεί καλύτερα εάν ε, μπορούν να αξιοποιηθούν αυτοί οι εργαζόμενοι σε διάφορους κλάδους. Και το τελευταίο, αυτοί οι εργαζόμενοι, οι κινητικοί εργαζόμενοι με βάση τις, ε, τους υπολογιστές. Αυτό δεν αφορά κλάδους αλλά συγκεκριμένα καθήκοντα. Το καθήκον πρέπει να επιτρέπει να εκτελεστεί ε, μέσω τεχνολογίας από το σπίτι σου, να μην χρειάζεται να πας στον τόπο εργασίας. Αν πρέπει να βοηθήσεις ας πούμε στην λιανική πώληση ή αν είσαι κομωτής, πρέπει να πας εκεί. Ή αν είσαι σερβιτόρος. Δεν μπορεί να είσαι από το σπίτι σου σερβιτόρος. Αυτό διαπιστώσαμε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ανεξάρτητα του κλάδου, είναι κυρίως ε, υπεύθυνοι διαχείρισης που μπορούν να μετακινούνται ή είναι εργασία με βάση υψηλό επίπεδο γνώσης σε μια διαφημιστική εταιρεία για παράδειγμα. Αυτή η δημιουργική εργαζόμενοι, αυτοί που αποφασίζουν τα συνθήματα των εκστρατιών. Δεν χρειάζεται να είναι επιτόπου. Επίσης σε μια εταιρεία ε, που ε, κάνει μετακομίσεις ε, ο προγραμματισμός του ποιος, ποιος οδηγός θα κάνει το οτιδήποτε θα αναλάβει την οποιαδήποτε μετακίνηση μπορεί να γίνει και από το σπίτι. Σας ευχαριστώ. Μια σύντομη ερώτηση και μια σύντομη απάντηση, κυρία Μορβάη. Πραγματικά η τελευταία ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Μία θεωρητική ερώτηση ήθελα να σας κάνω για να το διευκρινίσουμε. Ο στόχος της ε, απασχόλησης πέρα πολλών ε, άλλων ευγενών σκοπών είναι να μπορεί να ζήσει κανείς από τη δουλειά για να συντηρήσει τον εαυτό του, την οικογένειά του. Μου φαίνεται ότι οι άτυπες αυτές μορφές απασχόλησης, όπως για παράδειγμα να κάθεται κανείς στο σπίτι του και να περιμένει το τηλέφωνο του εκάστοτε εργοδότη και να σταυρώνει τα δάχτυλά του, και να κάνει και την προσευχή του, αυτές οι εργασιακές σχέσεις δεν αρκούν για να ζήσει κανείς. Συμφωνείτε με αυτή την αξιολόγησή μου. Και κατά δεύτερον, αυτές οι νέες εργασιακές σχέσεις δεν ε, μπορούν να τύχουν χρήσεων, ιδιαίτερα στα νέα κρατημέλη. Κατά τρίτον, η κυρία Μάκιντάιρ μίλησε για το πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να εφαρμόσουμε αυτούς τους διάφορους τρόπους απασχόλησης. Φαίνεται οι γυναίκες ε, από ένα ορισμένο κοινωνικό επίπεδο μπορεί να αποφασίσουν κάποια στιγμή να ε, δουλέψουν δύο-τρει εβδομάδε ε, για να βγάλουν ένα χαρτζελίκι, αλλά δεν υποχρεούνται να ζήσουν από αυτή τη μισθό. Ποιε είναι λοιπόν οι διαφορέ ό,τι αφορά τι άτυπε μορφέ εργασία μεταξύ νέων και παλαιών κρατών μελών, η απάντηση. Σα ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Και οι δύο ερωτήσει ε, είναι πάρα πολύ δύσκολε να απαντηθούν σε ό,τι αφορά τι νέε μορφέ απασχόληση εν γέννη, γιατί είναι τόσο ετερογενείς αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης που δεν θα μπορούσε κανείς να απαντήσει αρνητικά ή καταφατικά για όλες αυτές τις μορφές. Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα, σε ό,τι αφορά τις αποδοχές. Για, το, για τις πιο πολλές μορφές νέας απασχόλησης δεν είναι τόσο διαφορετικό, δεν είναι τόσο προβληματικό το θέμα αυτό, γιατί δεν είναι τόσο το διαφορετικό το επίπεδο αποδοχών. Αλλά σε κάποιες μορφές υπάρχει το ζήτημα αυτό. Και εδώ πέρα απομακρυνόμαστε από το να έχει κανείς ενδεχομένω μια σωστή δουλειά και μιλάμε σε πιο πολύ για ανάθεση έργων. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται το πρόβλημα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, την απασχόληση σε επιφυλακή, όπου κανείς λαμβάνει την εντολή το, για την απασχόληση, για τη δουλειά μία ώρα πριν. Έχει κανείς δηλαδή τις υποχρεώσεις, αλλά δεν μπορεί και να ζήσει παράλληλα από τη δουλειά αυτή. Και σε ό,τι αφορά το crowd employment, σε ό,τι αφορά δηλαδή στατιστικά στοιχεία για το ποιο είναι το εισόδημα των ατόμων αυτών. Και σε κάποιες περιπτώσεις μιλάμε για λεπτά του ευρώ. Αν δεν μπορεί κανείς λοιπόν να συγκεντρώσει πολλές τέτοιες ε, συμβάσεις, δεν μπορεί να ζήσει, ναι. Το κίνδυνο εκμετάλλευσης, ναι. Για τις μορφές εκείνες όπου η ευελιξία προβλέπεται μόνο για τον εργοδότη και υπερβολικά μεγάλη ευελιξία για τον εργαζόμενο και πάλι υπάρχει κάποιος κίνδυνος και εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας είτε από νομικής άποψης μεσολογικών συμβάσεων να υπάρχει πιο αυστηρή παρακολούθηση. Ναι, θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει. Δεν πιστεύουμε. Δεν βρήκαμε ιδιαίτερε διαφορέ μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών. Θα υπέθετα λοιπόν ότι το δυναμικό είναι το ίδιο παντού. Όπου υπάρχει ανάγκη και όπου δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος κατάχρηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μάντλ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Έγινε σήμερα μία συνεδρίαση σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ευελιξίας και καλύψαμε πολύ ενδιαφέροντες κλάδους και τομείς. Θα ήθελα μόνο να υπενθυμίσω στην Επιτροπή ότι η Eurofund στην οποία και εργάζεστε είναι δική μας, δικός μας οργανισμός οργανισμός απασχόλησης. Και η Επιτροπή μας πάντα έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, να σας ζητήσει νέα δεδομένα, νέες ε, μελέτες. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, χρήσιμο αυτό, το αποδείξατε άλλωστε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα γίνει 1η και 2η Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ.